Uh, uh, Καλημέρα σα. Έχουν έρθει εδώ οι κυριότεροι αρμόδιοι για το θέμα των επαγγελματικών προσόντων και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δεύτερη μας συνεδρία της εβδομάδας. Τις ανακοινώσεις μου τις έκανα χθες. Σήμερα θα σας πω στις 10 τα αποτελέσματα των συντονιστών που και θα έρθουν οι περισσότεροι για την ψηφοφορία. Λοιπόν, αρχίζουμε με μια ανταλλαγή απόψεων με την εισηγήτρια κυρία Μακκλάρκιν για έκθεση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. την ευχαριστώ και για το έγγραφο εργασίας της που είναι πολύ σημαντικό ως βάση για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων καθώς και τους σκιώδεις Ρεκρίκ, Βανούρε, ο κύριος Κρόιτσμαν νομίζω αντικαθιστά κάποιον και τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Επίσης καλωσορίζω τον κύριο Γιούργεν Τίτσερ που κάπου κρύβεται εκεί πίσω αλλά είναι ο υπεύθυνο από την Κομισιόν για αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ επίσης όλους που όσους λάβατε μέρος στην μικρή ομάδα ή επιτροπή ανάλυσης που κάναμε κατά την προπαρασκευή αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης. Αναμένω λοιπόν με ανυπομονησία αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με μεγάλη ειδονή δίνω το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και όλους εσάς που ήρθατε τόσο νωρίς. θα παραμείνω αυστηρά στο κείμενό μου το έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει στην ομάδα εργασίας, την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν έκανε και μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης που έκανε φέτος. Αυτά όμως δεν τα ανέφερα στο έγγραφο εργασίας γιατί δεν πρόλαβα. Κατανοείτε, ελπίζω, εδώ είναι ένα πρώτο έγγραφο, θα τα περιλάβω αργότερα. Κατά τη διαδικασία συλλογής ιδεών εδώ, θέλησα να δω τα συμπεράσματα διαφόρων διαβουλεύσεων και ομάδων εργασίας της Κομισιόν με τους ενδιαφερόμενους που με βοήθησαν πάρα πολύ για να καταλάβω ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Και ευχαριστώ την Κομισιόν και τα μέλη αυτά, τα κράτη-μέλη που μας βοήθησαν έτσι να καταλάβουμε κάπως περισσότερο τη λογική ορισμένων από αυτές τις προτάσεις. Βεβαίως πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων για να προσπαθήσουμε η οδηγία αυτή να γίνει πιο αποτελεσματική για όλους και όλες. Στόχος είναι να, καθοριστεί, να καθοριστούν οι κύριες προτεραιότητες για όπου μπορεί να χρειάζεται συγχρονισμός. Φυσικά είμαι πρόθυμη να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών και των υπολείπων συναδέλφων για να δω αν χρειάζεται περισσότερη αποσαφήνιση ορισμένων θεμάτων. Όπως λέει και από την εισαγωγή, η παροχή υπηρεσιών ε, σε άλλο κράτος μέλος είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον καθορισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα πρώτα σχετικά μέτρα ήταν η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική κινητικότητα και να υπάρχουν πιο ευέλικτες αγορές εργασίας με τον καθορι... μέσω του καθορισμού ομοιόμορφων διαδικασιών αναγνώρισης των προσόντων για να υπάρχει όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο χορηγής υπηρεσιών και προστασίας των καταναλωτών και καταναλωτριών. Αυτό το επιτυγχάνει η πρόταση γιατί υπήρξαν 171 απαντήσεις σε ερωτήματα που έθεσε η Κομισιόν ε, επαγγελματικοί οργανισμοί και απλοί πολίτες έτσι ώστε το σύστημα για την αναγνώριση να είναι, των προσόντων να είναι αποτελεσματικό και ρεαλιστικό. Υπάρχουν όμως ακόμη τομείς όπου τα κράτη-μέλη και οι επαγγελματίες ζητούν αλλαγές στις προτάσεις αυτές, πράγμα το οποίο θα συζητήσω αργότερα άλλη φορά σχεδόν χίλιοι εκπρόσωποι αρχών και 460 επαγγελματιών εξέτασαν την οδηγία και διαπίστωσαν ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν μετέφεραν σωστά ή και καθόλου την οδηγία. Άλλες υπηρεσίες όπως το Solvit ε, κατέληξαν ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην ισίουσα διαδικασία αναγνώριση ε, των προσόντων πράγμα για το οποίο έγιναν πολλά επίσημα παράπονα για τη δημιουργία διαγραφειοκρατικών φραγμών ή αγνία των βασικών πληροφοριών που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πού να αποταθούν. Πράγμα το οποίο μας οδήγησε να καταλήξουμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπιστοσύνης. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη παραπονεθεί και οι επαγγελματίες επίσης ότι δεν είναι διαφανείς οι διαδικασίες. Στην θεώρηση της οδηγίας αυτής θα πρέπει λοιπόν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αν τα λεγόμενα single points of contact μπορούν να βοηθήσουν τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επαφή με το κοινό και διάλογος με τις αρμόδιες αρχές. Η πρόταση της Κομισιόν τονίζει ότι είναι σημαντικό σε κάθε χώρα μέλος να υπάρχει ένα σταθερό και γνωστό εγνωσμένο σημείο επαφής με το κοινό. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα συμπληρωθεί η διαδικασία αυτή ηλεκτρονικά να μπορεί να συμπληρωθεί online Μερικές από τις διατάξεις της οδηγίας αυτής είχαν πρωτογραφτεί πριν από 30 χρόνια και επομένω χρειάζεται εξυγχρονισμός με διαβούλευση με το αρμόδια επαγγελματικά σώματα και οργανισμούς. Η Κομισιόν πάντως θεωρεί ότι της κατεξουσιοδότηση πράξη ω μια μέθοδο η οποία θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αγνοήσει τη, τη μέθοδο αυτήν. Άλλα συγκεκριμένα σημεία της οδηγίας έχουν ε, τύχει ιδιαίτερη προσοχής όπως η επαγγελματική κάρτα. Υπήρξαν ορισμένα πειραματικά ή πιλωτικά προγράμματα όπως για την European Engineers Association με την κάρτα του μηχανικού που χορηγούσε αυτή και η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτή η επαγγελματική κάρτα μπορεί να διευκολύνει τα πράγματα, να τα απλοποιήσει και να τα επιταχύνει ώστε να υπάρχει περισσότερη κινητικότητα των επαγγελματιών. Στο βήμα της ενιαίας αγοράς που θα οργανωθεί αργότερα φέτος θα τεθούν ξανά όλα αυτά καθώς και το θέμα της ευθύνης του κόστους και τα λοιπά για το θέμα αυτό της επαγγελματικής κάρτας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία αξιόπιστη αξιολόγηση με βάση στοιχεία από την πραγματική αγορά. Βέβαια πρέπει να είναι εθελοντική η χορήγηση αυτή της κάρτας η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες συγκεκριμένων επαγγελμάτων και να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία. Πρέπει να σκεφτούμε πολλά θέματα. Τι θα προσφέρει αυτό στους καταναλωτές, καταναλώτριες και επαγγελματίες. Τι πληροφορίες πρέπει να περιέχει, να αναφέρει, τι προστασία θα χορηγεί και το κυριότερο ίσως πώς θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και έγκρισης της κάρτας αυτής. Περιμένουμε βέβαια και τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια αξία έχει ή θα έχει αυτή η επαγγελματική κάρτα πριν να κρίνουμε τελικά. Αυτό φυσικά αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για την εσωτερική αγορά γενικότερα, το λεγόμενο IMI, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να υπάρχει καλύτερη διάδοση των πληροφοριών μεταξύ επαγγελμάτων και θα έπρεπε να μπορεί να ταυτίζει περιπτώσεις παραβίασης του δικαίου ιδιαίτερα ως προς τα επαγγέλματα που αφορούν την υγεία να υπάρχει ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας θα το πράττουν υπεύθυνα η έννοια της μερικής πρόσβασης είναι κάτι το οποίο και αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών. Η διαβούλευση που προβλέπεται δεν έχει εγκριθεί σε μεγάλο συστηματικό βαθμό μέχρι τώρα από τα κράτη-μέλη γιατί το πρόβλημα είναι πώς θα μπορούσε κανείς να ελέγξει την εφαρμογή του συστήματος. Η προσωρινή κινητικότητα που προβλέπει η οδηγία του 2005 επιτρέπει ένα πιο ευέλικτο σύστημα για τους επαγγελματίες τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και διευκολύνει την επιλογή του καταναλωτή και της καταναλωτρίας. αλλά υπάρχουν και εκεί προβλήματα που ενέφεραν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλες οι ενδιαφερόμενες και για την κινητικότητα και για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τη δημόσια υγεία. Η οδηγία λοιπόν δεν προέβλεπε ακριβώς πότε ακριβώς και για πόσο χρόνο θα έπρεπε, θα έχουν το δικαίωμα όσοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα να χωρικούν τις υπηρεσίες τους. Τέλος υπάρχει και το θέμα των γλωσσών, πολύ αμφιλεγόμενο, πάρα πολύ αμφιλεγόμενο. Ε, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Πρέπει οι επαγγελματίες να έχουν και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για να εργαστούν σε μια άλλη χώρα από τη δική τους γιατί διαπιστώθηκε ότι η οδηγία δεν ήταν πολύ σαφής ως προς το τι μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη-μέλη για να ελέγξουν τα επαγγελματικά προσόντα των επαγγελματιών. Στην πράσινη βίβλο της Οικομισιόν λέει ότι μπορεί μεμονωμένα κατά περίπτωση να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορεί το πρόβλημα να λυθεί πιο σφαιρικά μήπως πρέπει να υπάρξει κανένα νέο στοιχείο, καμία νέα διάταξη ρήτρα στην οδηγία για να διασφαλίζει τον έλεγχο των, γλωσσικών προσόντων για να μην υπάρχει και γλωσσικό εμπόδιο στη χορήγηση αυτών των υπηρεσιών. Σίγουρα θα καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσα να συζητήσω πολύ περισσότερο ορισμένα συγκεκριμένα θέματα, αλλά θέλησα να περιοριστώ σε αυτά που έθιξε η ίδια η Κομισιόν. Συνεδριάζω, συναντιέμαι με τους σκιώδεις σήμερα και αν κανείς ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα παρακαλώ να μου το πει τώρα για να τα πω και εγώ στους σκιώδεις. Χρονοδιάγραμμα, η, η έκθεση θα εξεταστεί στις 27 Ιουλίου και μετά τις διακοπές στις 30 Αυγούστου δεν ξέρω αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί, θα γίνει μετά μία βιντεοδιάσκεψη στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 17 Οκτωβρίου τελική έγκριση από την Επιτροπή. Επομένως, η αναθεώρηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα είναι ένα από τα κλειδιά για τη διασφάλιση της κινητικότητας στην εσωτερική αγορά. Πρέπει να ακούσουμε τα προβλήματα που έχουν να μας αναφέρουν οι επαγγελματίες για να διασφαλίσουμε αυτή την ενισχυμένη κινητικότητα. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε επίση και την ποιότητα των χορηγουμένων υπηρεσιών καθώ και όσον αφορά τα υγειονομικά, την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σφαιρική παρουσίαση. Εντοπίσατε τα σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε η 30... When we plan to, uh, to have a look at your draft report, um, uh, so that will be a... Ε, επιβεβαιώνω την 30 Αυγούστου, όπως είπατε. Ε, θα ξεκινήσουμε την κυρία Λεγκρίπ για σχόλια. Oui, merci, monsieur le, le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακκλάρκιν για την εξαιρετική της δουλειά. Και δεν είναι μονοτυπικές αυτές οι ευχαριστίες, πράγματι θέτει τα σωστά ερωτήματα. Το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων είναι κρίσιμο για το ευρωπαϊκό ιδεώδες και για την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο κύριος ο καθητής Μόντι στην έκθεσή του υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη να επεκτείνουμε την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων, ζήτησε να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αναγνώριση των διπλωμάτων, ενδεχομένως και με ένα ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης των επαγγελματικών προσόντων. Και ο Αλέν Λαμασούρ σε μια δική του έκθεση ε, είχε αναφέρει ότι για την Ευρώπη των πολιτών χρειάζεται να λυθούν τα προβλήματα της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων και προσόντων. Ε, η απουσία πλήρους και εύκολης αναγνώρισης ε, ακύρωνε ένα τμήμα της, ακυρώνει ένα τμήμα της Ευρώπης των πολιτών την οποία τόσο πολύ επιθυμούμε. Θα εξετάσουμε λοιπόν σήμερα την έκθεση αυτή γνωρίζοντας ότι ε, η αναγνώριση των παραγγελματών προσόντων είναι ένας από τους 12 μοχλούς της εσωτερικής αγοράς από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τη βάση, ως βάση την πράσινη βίβλο. Λοιπόν, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να ιδωθεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Από την επαγγελματική πλευρά βέβαια, από μια προφανώς, οι επαγγελματίες είναι οι πιο ενδιαφερόμενοι, θέλουν να χαίρουν της ελευθερίες κυκλοφορίας σε κράτη-μέλη εκτός του δικού τους. Επίσης θα πρέπει να τη δούμε από την πλευρά των ε, αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνε για την λήψη των αποφάσεων, ε, για την αναγνώριση την ίδια, αλλά πρέπει να την δούμε και από την πλευρά των ίδιων των χρηστών, των πολιτών και όλα αυτά με βάση κάποιες συγκεκριμένε αρχές. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη επαγγελματική κινητικότητα Δηλαδή αυτό είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να βρούμε τα μέσα έτσι ώστε να αυξηθεί η επαγγελματική κινητικότητα, να ξεπεράσουμε τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα. Περισσότερη λοιπόν κινητικότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα και απλούστευση στις διαδικασίες και μεγαλύτερη ασφάλεια για το κοινό, για τους καταναλωτές και ιδίως για τους ασθενείς, διότι ε, τα επαγγέλματα του, του κλάδου υγείας ε, είναι στο κέντρο της κινητικότητας. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων. Για τους επαγγελματίες είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η απλοποίηση. Πολύ συχνά είναι δυσχερέστατη ε, διαδικαστικά η μετακίνηση ενός εργαζόμενου σε άλλο κράτος, ε, μέλος, τεράστιες ε, καθυστερήσεις, ε, αδικαιολόγητες θα λέγαμε πολλές φορές. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε ένα αναλογικό σύστημα και αποτελεσματικό. Αναλογικό με την έννοια ότι χρειάζεται να εξισορροπήσουμε την ελευθερία κυκλοφορίας και εγκατάστασης με τις απαραίτητες εγγύσεις τα χέρια που θα πρέπει να δει το σύστημα στους καταναλωτές. Το θέμα της απλοποίησης ε, έχει σχέση με τον πολύ μεγάλο αριθμό 4.600 ε, συγκεκριμένων επαγγελμάτων ε, ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ο αριθμός αυτός να μειωθεί κατά πολύ λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη την πάντοτε τις ανάγκες που οδήγησαν στην ρύθμιση του κάθε επαγγέλματο. Αύξηση της κινητικότητας σημαίνει επίσης και αναθεώρηση των, της κατάρτισης για διάφορα επαγγέλματα. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε τα, τις ελάχιστους όρους ε, κατάρτισης και προσόντων για ορισμένα επαγγέλματα, ε, διότι πολλές φορές οι όροι αυτοί ε, είναι απερχιωμένοι και βασίζονται σε <clears throat> κριτήρια ε, που είχαν καθοριστεί πριν από μερικές δεκαετίες. Από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα συστήματα κατάρτισης σε πολλά κράτη-μέλη και θα πρέπει και εμείς να αναθεωρήσουμε, να επικαιροποιήσουμε τις απαιτήσει για τα προσόντα και την κατάρτιση ορισμένων επαγγελμάτων. Το θέμα κυρίως αφορά την ε, διαβίου επαγγελματική κατάρτιση ε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, για ορισμένα εργαλεία ε, τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Μακλάρκιν, θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής. Το σύστημα πληροφόρησης εσωτερικής αγοράς Νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνος, λειτουργεί ικανοποιητικά. Ε, χειρίζεται αρκετά γρήγορα τις ε, περιπτώσεις που του υποβάλλονται. Θα ασφαλώς θα πρέπει να το αναπτύξουμε, να το ενισχύσουμε, να του δώσουμε περισσότερα μέσα, οικονομικά και άλλα. Θα πρέπει να γίνει και πιο προορατικό σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα, κύριο, ένα κέριο σημείο, ε, κέριο σύστημα. Ε, το μηχανισμός προειδοποίησης ε, θα πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει θα πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό και αν ναι, αν πρέπει να είναι παρόμοιος με αυτόν της οδηγίας εσωτερικής αγοράς ή όχι κλπ. Ε, νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό του μηχανισμού. Ε, είναι απαραίτητο να προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ασθενών. Τώρα για την επαγγελματική κάρτα. Συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες και όλες τις ερωτήσεις που τίθενται σε ό,τι αφορά κυρίως ε, το κόστος, την αξιοπιστία, την πραγματική προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια τέτοια κάρτα. Ας δούμε τα αποτελέσματα των ε, πειραμάτων, των πιλωτικών προγραμμάτων, βέβαια, αλλά φαίνεται ότι πολλά επαγγέλματα ήδη έχουν ξεκινήσει, ε, ήδη μας ε, δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας μιας επαγγελματικής κάρτας που θα είναι και ένα διαβατήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ενδεχομένως πολλά από τα προβλήματα τα οποία θίγουμε ε, να έχουν ήδη λυθεί από ορισμένα ή πολλά επαγγέλματα. Διότι βλέπουμε ότι πολλά επαγγέλματα έχουν ήδη εκφράζουν ήδη τη βούληση να περάσουν ε, σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα τέτοιο εργαλείο. Βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του συστήματος, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει ε, να ε, ενημερώνουν το σύστημα αυτό τακτικά, να εξασφαλίζουν την, την ασφάλειά του Ενδεχομένω θα πρέπει οι κάρτες αυτές να είναι μαγνητικές κάρτες, ε, να μην είναι κάρτες σε χαρτί απλώς. Ε, τέτοια πράγματα εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, ε, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε γιατί είναι υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών και των πολιτών μας. Είναι, θα ήταν κάτι τέτοιο ένα απτό δείγμα ε, προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσε η Ευρώπη να δώσει στους πολίτες της. Για να εξασφαλίσει ότι η κινητικότητα και η ελευθερία εγκατάστασης ε, θα γίνεται με τρόπο ασφαλή. Με τις απαραίτητες βέβαια πάντοτε εγγυήσεις. Πάντως επαναλαμβάνω ορισμένα επαγγέλματα είναι ήδη έτοιμα. Ας προσπαθήσουμε πάντως ε, να μην είμαστε τελειομανείς, ε, προσπαθώντας να κατακτήσουμε την το... το τέλειο, ενδεχομένως δημιουργούμε περισσότερα εμπόδια στο δρόμο μας. Ε, αυτά ήταν τα σχόλιά μου. Νομίζω ότι το σχέδιο, το προσχέδιο αυτό θέτει τα σωστά ερωτήματα και περιμένουμε και τις άλλες νόμες. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπένιου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μακλάρκιν για τη δουλειά της, γιατί έθεσε τα σωστά θέματα και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα σε αυτό. Υπάρχουν ερωτήματα που τίθενται για αυτό το θέμα. Η συνάδελφος, η Γαλλίδα συνάδελφός μου είπε ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι τέλειο βέβαια, ιδίω για αυτό το θέμα που για μένα είναι θέμα κλειδί της θητείας μας και του μέλλοντος της Ευρώπης. Πολύ πολύπλοκο θέμα. Δεν θα τα λύσουμε σήμερα όλα τα προβλήματα βέβαια, ούτε και στα τέλη του Αυγού, ούτε και στο τέλος του Αυγούστου. Όμως είναι σημαντικό το θέμα διότι, όπως είπαν και άλλοι, 4.600 επαγγέλματα είναι νομικά διευθετημένα, υπάρχουν όμως πολλά που δεν είναι. Για το θέμα των επαγγελματικών προσόντων σημαίνει αφορά το 20% των θεμάτων που τίθενται στο Solvit. Είναι λοιπόν τεράστιο θέμα η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Πρέπει να καθοριστούν τα κατώτερα, για να το πω έτσι, προσόντα. Αυτό το ζητούν και οι επιχειρήσεις και είπατε και εσείς ότι είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες της αγοράς εργασίας αλλά και τους απλούς πολίτες ενδιαφέρει. Τι μας λένε οι πολίτες. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη αλλά και καλύτερη. Αλλιώς η κοινή γνώμη αν δεν μπορέσουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη τότε δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι το κόστος της είναι στην πραγματικότητα μια επένδυση για το μέλλον. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα αυτό με σαφή καθορισμό και χρονοδιαγραμμάτων μία γενιά, 10 χρόνια, 20 χρόνια, τότε θα έχουμε χάσει μια γενια δεκα χρονια εικοσι χρονια τοτε ευκαιρία για την οικοδόμηση της Ευρώπης και σε μερικά χρόνια λογικά τη στιγμή των ευρωεκλογών θα μας πούνε δεν δημιουργήσατε περισσότερη αλλά λιγότερη Ευρώπη. Και γι' αυτό ευχαριστώ και την Κομισιόν διότι όταν εξέτασα αυτό το θέμα το εξέτασα σε σύνδεση με, τις, με τα διαμεθοριακά και είχα πει ότι χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία για αυτά τα θέματα υγείας ιδίω περισσότερη κινητικότητα δεν έγινε τίποτα γιατί δεν υπήρξε καμιά φιλοδοξία. Τώρα όμως ευχαριστώ την Κομισιόν και τον εκπρόσωπό τη που θα μας μιλήσει λίγο γιατί βλέπω ότι είμαστε όλοι μαζί Κομισιόν και Κοινοβούλιο σύμφωνοι. Ελπίζω να μας ακολουθήσει και το Συμβούλιο σε αυτόν τον φιλόδοξο και ρεαλιστικό δρόμο που θα αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη απλοποίηση όπως ζητούν όλοι και όλες μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια και όλα αυτά είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί και μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργία των επαγγελματιών και των ασθενών και των καταναλωτών και καταναλωτριών και μεγαλύτερη προστασία πανενοσιακώς. Τεράστιο θέμα. Θα ταυτίσω τώρα ορισμένα προβλήματα κλειδιά που νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ ξανά την κυρία Μακλάρκιν για το πνεύμα με το οποίο εξέτασε το ανοιχτό πνεύμα αυτό το θέμα. Λοιπόν, τα σχόλια. Πρώτον για την εναρμόνιση των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν, να συνεργαστούν συνεχώς και σε μεγαλύτερο βάθος για να ορίσουν, να καθορίσουν από κοινού τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για ένα επάγγελμα. Επίσης όμως να διασφαλίσουν την συνεχή διαβίου μάθηση για να μπορεί κανείς να χορηγήσει υπηρεσίες στο εξωτερικό πρέπει να έχει και γλωσσικά προσόντα. Και θέλω να προσθεθεί εδώ το θέμα των επαγγελματικών εμπειριών, της επαγγελματικής εμπειρίας διότι ήδη υπάρχει κινητικότητα ακόμα και αν δεν βασίζεται σε νομισμένες διαδικασίες εκπαίδευσης. Βεβαίως θα χρειαστεί να κάνουμε και μία καλύτερη αξιολόγηση της διαδικασίας της Μπολόνιας όπου τα πράγματα δεν είναι τελείως αρνητικά αλλά ούτε και σαφέστατα για να μπορέσουμε έτσι να προσθέσουμε τη διαδικασία αυτή στα όσα ισχύουν εθνικώς και έτσι να δούμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε γιατί εδώ δεν συμφωνούν όλοι. Αφού λοιπόν μιλάμε για εναρμόνιση προσόντων και παιδείας πρέπει να μιλήσουμε και για την μερική πρόσβαση και για αντισταθμιστικά μέτρα για τη μερική πρόσβαση και για τη χορήγηση, προσωρινή χορήγηση υπηρεσιών ή χορήγηση προσωρινών υπηρεσιών πρέπει νομίζω να προσέξουμε ιδιαίτερα ένα πολύπλοκο θέμα γιατί μερική πρόσβαση μπορεί να σημαίνει και κατακαιρματισμό της αγοράς και εδώ πρέπει να προσέξουμε μήπως γίνει το αντίθετο από αυτό που θέλαμε Ο δεοντολογικός κώδικς καλός είναι αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή και στοχευμένη ανάλυση που να τον ξεπερνάει. Όσο για το σύστημα MIM ή IMI μάλλον και τον μηχανισμό προειδοποίησης και αυτά είναι απαραίτητα αλλά πρέπει να επεκταθούν. Τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταλαβαίνετε γι' αυτό. Λοιπόν, τα κοινά προγράμματα τώρα για αυτά τα θέματα εναρμόνισης η εφαρμογή τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας του 2005 απαιτεί συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών και των επαγγελματικών οργανώσεων. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει όντω ένα κοινό πρόγραμμα, κοινέ προτεραιότητε για προ στιγμή δεν συμβαίνει τίποτα. Ξέρετε ότι αυτό είναι το κύριο θέμα που με ενδιαφέρει. Το κύριο εργαλείο για καλύτερη κινητικότητα των επαγγελματιών, αν θέλουμε να διασφαλιστεί η διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια κτλ, είναι η κάρτα επαγγελματικής κινητικότητας εθελοντική βέβαια σε πρώτη φάση, ίσως και σε δεύτερη, ίσως και σε τρίτη. Αλλά είναι εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο πανενοσιακός, διότι ήδη υπάρχουν πειράματα, έχουν υπάρξει πειράματα που είχαν αποτελέσματα για τους κτηνιάτρους ας πούμε και γενικά για τον τομέα της υγείας. Την περασμένη εβδομάδα συζήτησαν το θέμα αυτό και οι λογιστέ. Δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αλλά και αυτοί θα ήθελαν αυτή την κάρτα. Επομένως οι εθνικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν, οι επαγγελματίες κάθε κλάδου πρέπει να καθορίσουν και το θέμα των διοριών του διάρκεια ισχύω της κάρτας τον τρόπο ενημέρωσής της, τον εμπιστευτικό ή μη χαρακτήρα των δεδομένων της. Και η κυρία Μακλάρκιν ρώτησε αν θα έπρεπε να είναι χάρτινη η κάρτα αυτή, αν θα έπρεπε να είναι ηλεκτρονική, αν θα έπρεπε να είναι πλαστική. Και νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να είναι ηλεκτρονική. Τίθεται και το θέμα του κόστους. Επειδή όμως εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτή η κάρτα, ξέρω ότι ο απλός πολίτης Ιδιαίτερα δε ο νέος και η νέα που ξέρει ότι το επαγγελματικό του μέλλον σημαίνει κινητικότητα και άρα χρειάζεται κάποιο διαβατήριο επαγγελματικό γνωρίζει ότι αυτή η επαγγελματική κάρτα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Οι 18 με 30 ετών θα χρειαστεί στο εξωτερικό να εργαστούν πάρα πολύ συχνά είναι σαν το θέμα της παιδείας σε κάθε χώρα. Η δική μου χώρα ξέρω έχει καθυστέρηση σε αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν πρόκειται για κόστος, είναι επένδυση, κοινωνική επένδυση, σημαντική επένδυση το εργαλείο αυτό. Το κόστος, το αρχικό κόστος θα αποσβεστεί εθελοντικά στην αρχή σε ορισμένα επαγγέλματα να γίνουν πειραματικά πιλωτικά προγράμματα και να δούμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος για 15-20 χρόνια. Δεν αυτά πατώμεθα. Αρχίζουμε απλώς κάτι, έναν δύσκολο δρόμο ακανθόδη. Αλλά πρέπει να στοχεύσουμε καλά του, να γνωρίζουμε ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι μας και ποιο είναι το κόστος για να, και να κάνουμε τακτικές επαληθεύσεις να έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκή έποψη της αγοράς των πολιτών και των επαγγελματιών. Και μόνο αν καταφέρουμε να συνεννοηθούμε επ' αυτού θα πετύχουν όλα αυτά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν συμφωνεί απολύτως μαζί μας, δεν, είναι και τόσο, δεν συμβαίνει και τόσο συχνά κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ως κοινοβουλευτικοί κάναμε τη δουλειά μας και μένει το θέμα των προσφυγών, δεν θα ήταν σωστό όλα να τα λύνει το δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πραγματικά ε, οξυδερκή παρουσίαση την οποία κάνατε. Αυτή τη φορά νομίζω ότι συζητάμε τα θέματα σε βάθος. Ε, πρέπει να πω ότι σήμερα ήμουν πάρα πολύ γενναιόδωρος ε, με τους ομιλητές γιατί έκρινα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχετε δυνατότητα να τοποθετείτε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στις 10 η ώρα ξεκινούν οι ψηφοφορίες. Επόμενος, ο κύριος Κρόιτσμαν θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Μπουζόη. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη ε, που δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στην ανταλλαγή απόψεων ε, καθαρά ε, για δικούς μου προσωπικούς λόγους ιατρικούς. Η εισήγηση αυτή είναι μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις έτσι ώστε να έχουμε μια έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη τη τις ε, Το έγγραφο εργασία ε, λαμβάνει υπόψη του πολλέ ε, προτεραιότητες. Υπάρχουν διάφορα σημεία ιδιαίτερη σημασία καταρχήν όσον αφορά την απλούστευση. Πράγματι υπάρχει περιθώριο απλούστευση. Η διαδικασία ενημέρωση για να πρέπει να συντονιστεί καλύτερα. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των πολιτών. Εξάλλου πρέπει να να εξετάσουμε και το σύστημα των δηλώσεων. Θα πρέπει να δούμε λιγάκι τη δυνατότητα οι δηλώσεις ε, να στέλνονται ε, online ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ε, δεν έχει κανένα νόημα να επιτρέπουμε στις ε, τοπικές αρχές ε, να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση ε, γιατί με τον τρόπο αυτό το θέμα καθίσταται περισσότερο περίπλοκο αποθαρρύνει τους Ευρωπαίους ως προς την κινητικότητα. Εξάλλου πρέπει να βρούμε λύσεις για να διευκολύνουμε τη μετανάστευση από μέλη που δεν έχουν προβεί σε ρυθμίσεις σε άλλα που έχουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις και αυτό, αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν μια σειρά επαγγελμάτων λύση είναι οι ρυθμίσει, οι κανονισμοί να ισχύουν μόνο εφόσον προστατεύουν το καταναλωτή, ε, την δημόσια υγεία ή ε, για άλλους αποχρόντες λόγους. Εξάλλου θα πρέπει να υπάρχει και το προαπαιτούμενο τη επαγγελματική εμπειρία, Σωστό αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί είναι η δυνατότητα να επιβάλλονται μέτρα αποζημίωσης. Ε, αυτά ε, στο πλαίσιο ε, των αποφάσεων που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι πρακτικές των κρατών μελών σε σχέση με τις αποζημιώσεις, τις επανορθώσεις ε, ε έχουν ήδη συζητηθεί. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια μέτρα επανόρθωσης που να αφορούν τις αρμόδιες αρχές η μερική πρόσβαση. Αυτό ε, μπορεί να ισχύει όταν τα καθήκοντα είναι ξεχωριστά, αλλά η μερική πρόσβαση δεν είναι καλή λύση για τέτοιου είδους επαγγέλματα όπου ο διοχωρισμός ε, είναι δυνατόν να λάβει χώρα ε, τη στιγμή που υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και για άλλους λόγους. Όσον αφορά την αναγνώριση, τα περισσότερα κράτη-μέλη απαιτούν να υπάρχει και μια πρακτική εφαρμογή, ελάχιστη πρακτική αφορμή Σωστά. Αυτό που έχει σημασία ε, είναι ότι δεν θα πρέπει απλά να δούμε τις ώρες ε, ή ε, το περιεχόμενο των μαθημάτων γιατί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Ένας μηχανισμός λοιπόν που θα επιτρέπει την προσαρμογή των ελάχιστων προδιαγραφών και θα δίνει τη δυνατότητα στην πραγματική αναγνώριση. Αυτό θα είναι πιο χρήσιμο. Εξάλλου για να υπάρχει αξιοπιστία στο σύστημα εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και των επαγγελματιών και των καταναλωτών, τα κράτη μελη πρέπει να διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη επικοινωνία όσον αφορά το περιεχόμενο της οδηγίας. Ο συνάδελφός μου πιστεύει ότι η χρήση του συστήματος IMI, του συστήματος ενημέρωσης εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ισχύει κυρίως όταν ο εφαρμοζόμενος, ο ενδιαφερόμενος έχει υποστεί καιρό σε ένα κράτο κράτος μέλος. Αυτό ισχύει κυρίως για τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, οι οποίοι πρέπει να αποκλείονται πράγμα που δεν είναι δυνατόν με την τρέχουσα νομοθεσία. Εξάλλου, η δημιουργία επαγγελματικών καρτών είναι κάτι το σημαντικό. Ο Κρίστιαν είναι υπέρ τη χρήση αυτών των καρτών στο βαθμό που προσφέρουν προστιθέμενη αξία για, για να μπορεί το σύστημα να είναι αποτελεσματικό πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Η χορήγηση επαγγελματική κάρτα θα πρέπει να χορηγείται κατά περίπτωση. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά στου μηχανικού, ε, ήδη υπάρχει εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, η οποία μοιάζει να είναι και θετική. Πριν λάβει αποφάσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Ο Κριστιαν συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι η κάρτα αυτή θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση αλλά εφόσον υπάρχει θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να τη δέχονται. Αλλιώς αφαλκιδεύεται η εξοπιστία της επαγγελματική αυτής κάρτας ευθύς εξ αρχής. Εξάλλου το σύστημα, η κάρτα μάλλον θα πρέπει να συνδέεται με το σύστημα ενημέρωσης εσωτερικής αγοράς, το IMI. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλώ να στείλετε ε, τις ευχές μας ε, για ταχύ ανάρρωση στον Κρίστιαν. Ε, Επόμενη, <clears throat> Κύριε Τούρινγκ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το έγγραφο εργασία. Είναι ένα πολύ καλό ε, σημείο κίνηση ε, για όλου μα. Νομίζω λοιπόν ότι επιτύχατε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που είναι σημαντικό, που είναι βεβαίω να βελτιωθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη, αφενό αυτό και αφετέρου την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων. Αυτό είναι ο στόχο. Νομίζω ότι στην αίθουσα όλοι συμφωνούν επ' αυτού. Εξάλλου ε, παρουσιάσατε και τα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται και τις προτεραιότητες όσον αφορούν ε, στην εφαρμογή, στην απλούστευση ε, θεμάτων υγείας και ασφάλειας. Ε, όταν θέσατε το θέμα για την επαγγελματική κάρτα, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στην ουσία αυτή τη κάρτα, δηλαδή πώ θα εφαρμόζεται αυτή η κάρτα. Και όπω είπατε και εσεί ε, προηγουμένω, όλα βεβαίω εξαρτώνται από το σύστημα που στηρίζει αυτή την κάρτα. Νομίζω πολύ σωστά υποβάλλεται αυτέ τις ερωτήσει και νομίζω οι σκιώδει ηγητέ θα πρέπει να προχωρήσουν ένα βήμα περισσότερο σε συνεργασία με την Κομισιόν για το πώ μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η κάρτα. Ε, και υπάρχουν και κάποια άλλα που θέλω να πω. Βέβαια σε πολλά καλύφθηκα. Θα πω μόνο ότι ε, πρέπει να αποδώσουμε δώσουμε λίγο μεγαλύτερη σημασία στα εξή. Πρώτον, να είμαστε περισσότερο ακριβείς όσον αφορά στη μερική πρόσβαση. Αυτό αφορά και άλλου ηγητέ. Ε, το αναφέρετε στο έγγραφο εργασία, αλλά δεν λέτε ακριβώ τι πρέπει ε, να γίνει με τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Τι πρέπει να γίνει στον τομέα τη υγεία. Πώ μπορούμε να επιλύσουμε τα εφιστάμενα προβλήματα. Κατόπιν, Όσον αφορά στους νέους απόφοιτους, νομίζω είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο έθεσε η ομάδα εργασίας. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους απόφοιτους αυτούς ε, να έχουν κινητικότητα, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορεί κανείς την πρώτη δουλειά να την αποκτήσει σε μια άλλη τρίτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε στον, στην αυτόματη αναγνώριση και αυτό πρέπει να το δούμε. Τέταρτον, αναφέρθηκα ήδη στην κάρτα. Πέμπτον, αφορά στη γλώσσα. Νομίζω αναφέρεται ένα κώδικα συμπεριφοράς ε, ως ένα μια δυνατότητα λύση, αλλά χρειαζόμαστε πιο αυστηρές διατάξει. Ε, Κυρίω όταν αυτό σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια. Δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρω αν βρήκα εγώ τι ε, σωστέ λύσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε. Ένα έκτο σημείο είναι το εξής. Έλαβα ε, πολλά μηνύματα από διάφορους επαγγελματίες και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Προσεκτικοί όταν τα προσόντα μια ομάδας επαγγελματιών δεν την χάνει αναγνώριση σε ένα κράτος μέλος. Είναι δύσκολο να υποσχεθούμε ότι ένα επάγγελμα θα συμπεριληφθεί στα ήδη αναγνωρισμένα, αλλά μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα. Το τελευταίο, ε, παιδεία σε σχέση με την εκπαίδευση. Συμφωνώ με την κυρία Μπένιου ότι χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία, ε, ελάχιστες ε, προδιαγραφές. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε ε, τα διαφορετικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αν όμως ε, θέλουμε κινητικότητα πρέπει να υπάρχει και μια ελάχιστη βάση πάνω στην οποία θα τη στηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι σε την Επιτροπή θα κάνουμε καλή δουλειά όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σκιώδης μας κυρία Σβέντσον, δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά θα ε, έρθει σε μια επόμενη συνεδρίαση να σχολιάσει όλα αυτά τα σημαντικά θέματα, τη γλώσσα, την επαγγελματική κάρτα και όλα αυτά. Οπότε οι απόψεις της ομάδας μας θα συμμεριθούν στην έκθεση. κυρία Βένσον θα έρθει σε επαφή με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για μια-δυο ακόμα παρεμβάσεις. Η κυρία Στάιρο. Κανείς άλλος. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ σχεδόν με όλα όσα ελέγχθησαν. Ιδιαίτερα για το θέμα της επαγγελματικής ε, κάρτας ίσω χρειάζεται πράγματι μια μελέτη επιπτώσεων. Να υπογραμμίσω επίση και το θέμα των γλωσσών και να θέσω το εξή ερώτημα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει εξετάσει πώ αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό των γλωσσών, ιδιαίτερα στον τομέα υγεία στα κράτη-μέλη. Γιατί ορισμένα κράτη-μέλη δείχνουν να ε, έχουν καλύτερα συστήματα από κάποιε άλλε. Τι χρησιμοποιούν διερμηνεί, τι κάνουν. Επίση, για το, για το ελάχιστο σύνολο προσόντων, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά με τα δοντιατρικά επαγγέλματα. Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένε χώρε. Κάποιο μπορεί να πάρει τον τίτλο του γιατρού και ταυτόχρονα ε, να του, να του δοθεί δυνατότητα να εργάζεται ως οδοντίατρο σε άλλα κράτη-μέλη σε άλλο κράτος μέλος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της υγείας στον τομέα του, το, της ασφάλισης τομέα της υγείας. Συνεπώς υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα ότι οι γιατροί εργάζονται ως οδοντίατροι. Ε, υπάρχουν τέτοιες, ε, μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό γιατί μου έχει καταγγελθεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για το πώ θα εξασφαλίσουμε την κινητικότητα, ασφαλώς, αλλά ταυτόχρονα πώς θα εγγυηθούμε για την ασφάλεια των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Styler. Right. Um, I don't see anybody else wanting the floor, um, so I'm going to invite teach it perhaps as well, but I'm very pleased to welcome you here and uh, to give you the floor. Ε, από, για την ε, Κομισιόν. Ο λόγος στην Κομισιόν. Ευχαριστώ την κυρία Συγγετρία. Τέσσερις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Όπως είπαν καταρχήν πολλοί ε, αρκετοί ευρωβουλευτές, η οδηγία αυτή αποτελεί προτεραιότητα και Εκτό από προτεραιότητα είναι και, αποτελεί και ένα χρονοδιάγραμμα, θέτει ένα χρονοδιάγραμμα σε όλου μα. και ευχαριστώ πάρα πολύ που όλοι σα δείχνετε την ε, επιθυμία να προχωρήσουμε γρήγορα. Να σα υπογραμμίσω επίση ότι το θέμα θα συζητηθεί στο τέλο Σεπτεμβρίου και από το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητα. Δεύτερη παρατήρηση για το θέμα των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, το αριθμού των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Το θέμα αυτό είναι περίπλοκο αυτό που ρωτήσαμε στην Πράσινη Βίβλο δεν έχει σχέση μόνο με τον αριθμό, αλλά και ε, έχει σχέση με το τι μπορεί να κάνει αυτή η οδηγία για να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε την Πράσινη Βίβλο. Κοιτάξτε τι προτείνει η Πράσινη Βίβλος άμεσα και έμεσα. Ε, για παράδειγμα, η ρυθμιζ... αναφέρεται στη ρυθμιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση. Οπότε εγώ κάνω ε, σύνδεση ανάμεσα σε αυτά δύο ζητήματα στην Πράσινη Βίβλο. Δεύτερον, για το IMI, το Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς. Το IMI δεν αναφέρεται αυτή τη στιγμή στην Οδηγία Επαγγελματικών Προσόντων. Στη συζητήση σας όμως ε, να το λαμβάνετε παρακαλώ ως δεδομένο γιατί λειτουργεί. Και μέχρι το 2000 και από το 2012 και μετά δεν θα καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο αριθμό ε, ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, αλλά όλα τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Αυτό το έχουν ήδη συμφωνήσει τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έρχομαι έτσι στην τέταρτη παρατήρησή μου, ε, που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα. Ας είμαστε σαφείς η Κομισιόν δεν επιθυμεί απλώ να υπάρχει μια ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα για να την ε, κυκλοφορεί κάποιο ε, στην τσέπη του και να έχει τη φωτογραφία του πάνω. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Η πράσινη βίβλος είναι, είναι πολύ σαφή αυτό το ζήτημα. Και ίσως θέλετε και εσείς να το σκεφτείτε. Εμείς συνδέουμε το σύστημα IMI με την υποστήριξη της επαγγελματικής κάρτας. Δηλαδή, το IMI χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε το κόστος του. Και υπάρχει, ακολουθείται και μια στρατηγική επέκταση του IMI, την οποία παρουσιάσαμε το Μάρτιο. Συνεπώς, το IMI θα μπορούσε να καλύψει τις επαγγελματικέ κάρτες. Δέστε αυτά τα δύο πράγματα μαζί, σε συνδυασμό. Δεν πιστεύω ότι το IMI από μόνο του αποτελεί βεβαλήση. Εμείς προτείναμε όσοι έχουν επαγγελματική κάρτα να αναγνωρίζονται αυτόματα, όχι σε τρεις μήνες, σε δύο εβδομάδες. Και αν κάποιος ζητήσει προσωρινή κινητικότητα, θα μπορούσε η αναγνώριση να γίνει σχεδόν χωρίς καθόλου γραφειοκρατία ή και χωρίς καθόλου. Η, τα εχέγγυα θα τα εξασφαλίζει το IMI. Τις εγγύης θα τις δίνει το IMI. Το IMI θεωρήστε το ως δεδομένο. Υπάρχει, λειτουργεί. Αν όμως στηριχτούμε μόνο στο IMI, ε, θα έχουμε κάνει ένα στρατηγικό λάθος. Γιατί, Γιατί το IMI είναι κάτι που ανάγκασε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Αλλά δεν έχουν πρόσβαση στο IMI ούτε οι πολίτε ούτε οι επαγγελματίε και δεν θέλουμε να έχουν πρόσβαση για να μην το υποσκάψουμε. Αλλά ε, ποια είναι τα ωφέλη τα οποία μπορεί να αντλήσει από το IMI ένα πολίτη. Ε, μπορεί κάποιο να έχει δικαιώματα πιο γρήγορη αναγνώριση επειδή τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του πιο γρήγορα. Ναι, υπό την προπόθεση ότι θα υιοθετήσουμε την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα. Αυτό θα είναι ο κοινό παρανομαστή πολλών επαγγελμάτων και αυτό έχουμε υπόψη μα ω όφελο του επαγγελματία και του πολίτη από το IMI, το οποίο θα υποστηρίζει την επαγγελματική αυτή κάρτα. Σκεφτείτε τα αυτά. Οι εμπειρογνώμονες θα συναντηθούν στην Κρακοβία στις αρχές Οκτωβρίου και εκεί θα συζητήσουμε και θα εκθέσουμε το πώ το IMI μπορεί να συνδυαστεί με μια ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα. Ευχαριστώ. Uh, uh, σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για το πώς ακριβώς η τεχνολογία και η συνεργασία μπορεί να μας ε, βοηθήσει. Ε, πράγματι, πολύ σωστό το όραμά σας σχετικά με την οδηγία που όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι μεγάλη σημασία και είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που εξετάζουμε. Πράγματι είναι μια οδηγία οξυδερκής όπως τη χαρακτήρισα. Ε, οι περισσότερες παρεμβάσεις σήμερα το πρωί ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Προφανώς ε, και τη εισηγήτριάς μας ε, που έθεσε ένα πολύ σωστό πλαίσιο. Αλλά βλέπετε πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα και βλέπετε ότι η δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα έχει αρχίσει να αποδίδει. Βλέπουμε πόσο οραματική είναι η προσέγγιση αυτής της Επιτροπής ε, νομίζω ότι αναφερθήκατε είδα στο χρονοδιάγραμμα, αλλά αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε πριν ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, ε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και για όλα αυτά που ακούστηκαν ε, σήμερα το πρωί. Ήσασταν όλα ιδιαίτερα ενημερωμένοι για το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι με την έκθεση αυτή θα προσθέσουμε κάτι, θα προκαλέσουμε μια βελτίωση, μια διαφοροποίηση. Μέχρι τώρα συνεργαστήκαμε και ε, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ε, το θέμα της κάρτας. Κοιτάξτε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το δίπλωμα οδηγού με φωτογραφία και όταν εγώ χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω το δίπλωμα οδήγησης ε, για άλλους λόγους πέρα από το να αποδείξω ότι είμαι οδηγός πρέπει να έχω και ένα σχετικό έγγραφο που να την πιστοποιεί. Δηλαδή η κάρτα από μόνη της δεν αρκεί για πιστοποίηση για άλλες περιπτώσεις. Μπορεί αυτό που λέτε για την επαγγελματική κάρτα να είναι η βέλτιστη λύση, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Βένιου, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό παράλληλα και με άλλα, όπως με την ε, οδηγία περί προστασία δεδομένων. Και τώρα είναι πλέον η ευκαιρία που μας ε, προσφέρεται ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σύστημα των προσόντων, έχοντας εξετάσει το σύστημα αυτό και κάτω από την προστασία των δεδομένων. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι να το χρονικό διάστημα για την ε, κατάθεση αιτήσεων ε, να ισχύει το σύστημα IMI, συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεμπάστιαν από τη Γραμματεία για τη βοήθεια που μου προσέφερε και ευχαριστώ πολύ και τους συμβούλους μου. Πάντως προσβλέπω στην συνέχιση συνεργασία με όλους σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς βέβαια προσβλέπουμε στο να γίνει αυτή η συζήτηση ξανά στις 30 ε, Αυγούστου. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ε, ημερομηνίες, οργανώνουμε μια ε, τηλεδιάσκεψη με την Επιτροπή του Bundestag στις 19 Σεπτεμβρίου. Θα ρυθμίσουμε όλα τα τεχνολογικά και όσον αφορά την έκθεση Μακάρθη, μετά έχοντας εξετάσει την έκθεσή της στις 30 Αυγούστου η διορία είναι 22 Σεπτεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών. Έχετε λοιπόν μεγάλο χρονικό περιθώριο για να τοποθετηθείτε. Μετά θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου και το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα ε, και θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά. Προχωράμε τώρα. Ε, πάμε στις ε, ψηφοφορίες πληροφορίες ε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα της ημέρησης διάταξης. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, ε, θέλω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις, γιατί εδώ έχουμε αρκετούς συναδέλφους παρόντες. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι σήμερα το απόγευμα ε, αλλάζει λιγάκι η ημερήσια διάταξη όσον αφορά στα θέματα που θα εξετάσουμε. Η κυρία Στάιλερ και η κυρία Βαντεκάμ συμφώνησαν να αλλάξουν τη σειρά ε, δηλαδή η κυρία Στάιλερ γύρω στις 5.30 θα παρουσιάσει την έκθεσή της και ο κύριος Βαντεκάμπ λίγο πριν από τις 6 ε, το απόγευμα. Ελπίζω να έχει φτάσει ο κύριος Βαντεκάμπ. Θα ήθελα σύντομα να σας ε, ενημερώσω για κάποιες σημαντικές αποφάσεις που έλαβαν χτες οι συντονιστές, κυρίως όσον αφορά την την ανάθεση εκθέσεων. Όπως ξέρετε όλα τα μέλη ε, παίρνουν τις αποφάσεις σε γραπτή μορφή μετά τις συνεδρίες των συντονιστών. Όσον αφορά όμως τις νέες εκθέσεις για τις οποίες θα αρχίσουμε να θα καταρχήν όσον αφορά την οδηγία ευρωπαϊκής τυποποίησης που είναι πολύ σημαντική, ε, θα πάει στην ΕΛΚ. Ο κύριος, η κυρία Κόμη, ε, η αντιπρόεδρος, θα λάβει αυτή την έκθεση. Τη συγχαίρω για αυτή την πολύ σημαντική ανάθεση. όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στους φιλελεύθερους, φιλελεύθερους ε, Κρόιτσμαν. Αυτές, ε, είναι οι δύο νομοθετικές προτάσεις που θα αρχίσουμε να εξετάζουμε και έχουμε και άλλες σημαντικές ε, γνωμοδοτήσεις. Χρήση φανών έργων, αυτό πηγαίνει στους φιλελεύθερους. Ο κανονισμός για την διατροφή ε, των νέων παιδιών στο ΕΛΚ, ε, η έκθεση για το ρόμι, για την περιαγωγή, ε, για αυτήν κάναμε μια σημαντική γνωμοδότηση τελευταία φορά ε, όσον αφορά ε, το scoreboard της ιστορικής αγοράς στο ΕΛΚ, τη στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών στους σοσιαλιστές. Αυτές είναι οι γνωμοδοτήσεις και μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις ε, δικαιώματα των ταξιδιωτών, φιλελεύθερη, έκθεση ανταγωνισμού στους συντηρητικούς, τρόφιμα στο ΕΛΚ, ανταγωνιστική κοινή αγορά ε, στην ομάδα των σοσιαλιστών, σταθεροποίηση της διαδικασίας Μπολόνιας. Ε, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και αυτή νομίζω μπορούμε να τη συνδυάσουμε με την έκθεση Μακλάκ. Ε, το πλαίσιο Corporate Governance, ΕΛΚ, Ιθαγένεια, Σοσιαλιστές και Πολιετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο φιλελεύθεροι. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές εργασίες ε, που πρέπει να γίνουν ε, πριν από σερινές διακοπές ή καντιά των διακοπών και προσβλέπω σε αποτελέσματα στην όπορ και κάποια άλλα θέματα που αφορούν όλα τα μέλη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη σημασία του Φόρουμ της κοινή Αγοράς. Ακρόαση θα οργανωθεί σήμερα το απόγευμα από την Πολωνική Προεδρία. Θα λάβει επίσης χώρα 2-4 Αυγούστου στην Κρακοβία. Μεταξύ άλλων ο κύριος Μπουζόη συμμετέχουν σε αυτή την ακρόαση. Έχουμε και ένα σχετικό πρόγραμμα. Ε, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει συμφωνήσει να πάει πλήρης αντιπροσωπεία σε, αυτή, σε αυτό το φόρουμ. Θα έχετε λοιπόν πολύ να ε, λάβετε μέρος σε αυτό το φόρουμ. Και δεύτερον, εξετάζουμε τη δυνατότητα επιπρόσθετης αποστολής στην Δανία εφέτος, γιατί έχουμε άδειε σε κάποιες θέσεις και θα σας ενημερώσω έγκαιρα ε, και θα το ακούσετε και στις αποφάσεις προτάσεις των συντονιστών αργότερα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Για σήμερα έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη αφορά την γνωμοδότηση για τους κινδύνους από μεγάλα ατυχήματα με επικίνδυνες ουσίες της κυρίας Χάνσλικ και ε, έχουμε εδώ την εισηγήτρια, την κυρία Και ε, Θέλετε να πείτε κάτι πριν από την ψηφοφορία. Κυρία Χάνσλικ, ε, η έκθεσή σας θα ψηφιστεί Έχετε να πείτε κάτι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, συζητούσαμε μερικά θέματα εδώ με τον Άντρες. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους όλους ηγητές για την εξαιρετική συνεργασία τους. Ελπίζω ότι η έκθεσή μου αντικατοπτρίζει τα, τα σχόλια και τις νόμες όλων των συναδέλφων. Οπότε ε, ζητώ να την υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Right. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Αν χρειαστούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα κοιτάξουμε το σύστημα. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε ε, ότι όλοι είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία. Έχουμε ε, αρκετό αριθμό συμμετεχόντων. Ξεκινάμε με, το 20, με την τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της κυρία Χάνσλικ και πάλι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 της κυρίας Χάνσλικ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Της ηγετρίας υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, γλωσσική, τροπολογία 11, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12, της ηγετρίας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, καταπίπτει. 26, της κυρίας Παρβανόβα, ως προσθήκη, νομίζω έχει σύμφωνη με τις ηγετρίας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 της ηγήτριας υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Uh, the votes... Ψηφοφορία λίγη. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ 10 κατά. Τροπολογία ε, περνάμε στην 28 κατευθείαν. Ε, Γκόγεν Πέρες, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της ηγήτριας, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 της κυρίας Παρβανόβα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 30 της κυρίας Παρβανόβα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 31 ως προσθήκη της κυρίας Ιργκοϊν Πέρεθ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 έχει αποσυρθεί. 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της ηγήτριας. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Γλωσσικής φύσεως. Πέραμε στη 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης. Στο παράρτημα 1 έχουν αποσυρθεί αρκετές τροπολογίες. Περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Κατά. Εγκρίνεται. Αυτό ήταν προστίκη. Τροπολογία 4. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της νομοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ομοφωνία. 32 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Χάντσλικ. Θα υποστηρίξετε τις τροπολογίες μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Περνάμε σε την επόμενη νομοδότηση για την Επιτροπή Βιομηχανίας για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο έρευνας και, και καινοτομίας. Συγγετρία κυρία Κόμη. Λάρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πριν περάσουμε στην ε, ψηφοφορία των τροπολογιών, ε, θα ήθελα πολύ σύντομο, σύντομα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία με όλους τους σκιοδησηγητές και τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη δουλειά ως έλαβε χώρα. Ε, λάβαμε υπόψη μα ε, τι ε, τροπολογίε και τι ε, συμβαστικέ προτάσει. Κατατέθηκαν πάρα πολλέ τροπολογίε και αυτό φαντάζομαι για το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κατά τη διάρκεια τη ψηφορία είχαμε και μια προφορική τροπολογία, την 29, την οποία και θα σα διαβάσω κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω όλου γιατί ήταν πράγματι μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και σε σχέση με αυτά τα οποία μα είπε η Επιτροπή Βιομηχανία. Σας ευχαριστούμε πολύ και πράγματι συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική πρόταση. Ας πάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπέρτατα αποχές εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα... σε τρία που αφορούν το ένα. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι οι τροπολογίες Γκρέκ και Ράπτη. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνονται 18 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία υπερθμών 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποθές, εγκρίνεται. Η, τροπολογία 6. Η 6 παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. 14 κατά. Η 7 του κυρίου Γκρέκ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται. Εγκρίνεται αυτή. Η 9 του κυρίου Φόξ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 8 ε, Μπιζόη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 Fox και εγώ και του υποφαινόμενου υπέρ κατά γκρίνεται η 13 του κυρίου Φόξ υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ αν και νομίζω απορρίφθηκε υπέρ κατά απορρίπτεται η 15 της κυρίας Ράπτη υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνεται κατόπιν του καταπίπτει 14. Πάμε τώρα στην σημαντική πρόταση 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν πάμε τώρα στην 19 του κυρίου Γκρέκ υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 20 της κυρίας Ράπτη αρχίζει ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 20. Έκλεισε. Απορρίπτηκε. απορρίπτηται. 19 ε, και 15 υπέρ. Η 3 συμβαστική υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Η 22 της κυρίας Ράπτη υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική υπαριθμών 4. Εδώ έχουμε ψηφορία κατά τμήματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ε, θα ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου χωρίς τις λέξεις ε, από νέους και γυναίκες επιχειρηματίες υπέρ, κατά, αποχές, ε, συγγνώμη, εγκρίνεται. Και μετά πάμε στο υπόλοιπο τμήμα υπέρ, κατά. Εγκρίνεται και αυτό. Νομίζω τώρα πάμε πιο κάτω στην τροπολογία υπεριθμών 29 με ε, προφορική τροπολογία, η οποία αναφέρεται όμως ε, ε, στο έγγραφο μπροστά μας Νομίζω είναι σαφέ, δεν χρειάζεται. Θέλετε, κυρία Κόμη, να το σχολιάσετε. Όχι, η τροπολογία αναφέρεται με πλάγια γράμματα υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Καταπίπτει 29. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε για την 31. Υπέρ παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 31. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Στο όριο, αλλά απορρίφθηκε. Η 32. Μπαλτσίτης, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίνεται. Η 5. Γκρέκ και Ράπτη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 5. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 18 κατά, 16 υπέρ. Η 10 Μπουζόη. Ψηφίζουμε για τη 10 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε με μία ψήφο. Κάτι δεν έγινε, κάποιος δεν ψήφισε. Απορρίφθηκε. 17, ε, με 16. Και πάμε τώρα στην παράγραφο 8, η 36, Βερνιό. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 36. Έκλεισε. Απορρίφθηκε. Η 34, Γκρέκ, υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 39, υπέρ. Κατά. Επίσης εγκρίθηκε. 41 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 41. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 21 με 13. 43 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μισό λεπτό, οριακό το αποτέλεσμα. Μάλλον έκλεισε, έκλεισε η ψηφορία. Απορρίφθηκε επίση. Ναι, 17 με 17, οριακό. 38 του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Επίση οριακό το αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε 45 υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίθηκε. 48 υπέρ κατά, επίσης εγκρίθηκε. Τώρα λοιπόν ε, ψηφίζουμε για το σύνολο του σχέδιου ε, ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφορία. Και έκλεισε. Και εγκρίθηκε το σχέδιο ψηφίσματος με 33 υπέρ, ε, μία εποχή. Συγχαρητήρια κυρία Κόμη. Και Θέλουμε να βασιζόμαστε σε εσά ε, ότι θα υπερασπιστείτε τη θέση μας στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Τώρα λοιπόν ελπίζω να παραμείνετε για το επόμενο θέμα γιατί έχουμε μια σημαντική παρουσίαση και αμέσως μετά, ναι, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση ε, από τον κύριο Ροσφόρ για το σχέδιο γνωμοδότησής του που αφορά την εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Ε, αυτά τα δύο θα τα συνδυάσουμε, τη μελέτη και την ε, έρευνα του κυρίου Ροσφόρ. Έτσι λοιπόν ε, πρώτα ο ίδιος θα σχολιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης αν κάποιος δεν θέλει να φύγει, ε, θα είχε στην καλοσύνη να φύγει ήσυχα από την αίθουσα, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Πρόκειται για μία μελέτη, ε, την οποία αναθέσαμε εμείς για την διασυνοριακή εναλλακτική επίλυση διαφορών ε, για να εξετάσουμε λιγάκι το θέμα αυτό στα κρατημέλη, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και θελήσαμε να αποκτήσουμε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρόκειται για ε, την προετοιμασία μιας μελέτης ε, που γνωρίζουμε ότι θα μας στείλει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξάλλου νομίζω ότι έχουμε εδώ ε, και μέλη από την μάλλον εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ, την κυρία Ρουίζο, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος αυτού για να ακούσει ε, την παρουσίαση και θα κληθεί να μιλήσει αργότερα. Είναι λοιπόν μια μελέτη ε, που έγινε από την Civic Consulting, από αυτή την εταιρεία. Έχετε τις ε, διαφάνειες φωτοτυπίες των διαφανειών και νομίζω ο κύριος Αλεβελτ που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρεία. ο κύριος Άλεβελτ έχει κάνει πολλές μελέτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για αυτή την Επιτροπή. Ο κύριος Άλεβερτ θα παρουσιάσει, θα κάνει την παρουσίαση. Έχουμε επίσης την κυρία Νατιγκάλ, τον κύριο Βαν και την κυρία Φερμπέκε από την Civic Consulting. Όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση. Και θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Άλεβελτ για να κάνει την παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Θέλετε τα φώτα αναμένα ή σβησμένα για τις διαφάνειες. Για να δω. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Η παρουσίαση είναι σε τρία τμήματα. Η νομική ανάλυση τριών νομοθετικών εργαλείων και μετά τα συμπεράσματα για την ΕΕΔ. Ο πρώτος παρουσιαστής. Η πρώτη παρουσιάστρια μάλλον. Ευχαριστώ. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών τι εννοεί επίλυση διαφορών εκτός δικαστηρίων με τη χρήση νενομισμένων μηχανισμών συμπεφωνημένων, προσυμπεφωνημένων. Γενικά στην Ένωση έχουμε ταυτίσει περίπου 750 μηχανισμούς ΕΕΔ. 470 έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν και βασίζονται σε διάφορες οδηγίες. Αυτοί οι μηχανισμοί ε, ε, δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους αλλά έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να τις ταξινομήσουμε. Είναι ιδιωτικά, δημόσια, βασίζονται στον ιδρυτή τους, στη χρηματοδότηση τους ή τα διαφοροποιούμε με το κατά πόσον συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, αν είναι δεσμευτικά ή όχι τα αποτελέσματα, αν είναι εθνικά ή υπερεθνικά και αν καλύπτουν έναν ή περισσότερους τομείς. Έχουμε ταυτίσει λοιπόν μια τάση που αυξάνεται χρήσης των εναλλακτικών αυτών μηχανισμών. Το 2008 οι περιπτώσεις ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο. Δεν μπορώ να ταυτίσω ακριβώς τους λόγους για αυτή την ανωδική τάση. Ίσως είναι γιατί είναι πιο διαθέσιμα αυτά τα προγράμματα, οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Πρέπει να τονίσουμε ότι η χρήση του ΕΕΔ διαφέρει κατά πολύ ανάλογα με τις χώρες. Εδώ με τα διαφορετικά χρώματα βλέπετε ότι τα πιο σκούρα χρώματα σημαίνουν περισσότερη χρήση τους και τα ελαφρύτερα, τα πιο ανοιχτά, μικρότερη. Το Βέλγιο φαίνεται να χρησιμοποιεί τις περισσότερες 4,73 περιπτώσεις ανά χίλιους κατοίκους και ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο και στο αντίθετο άκρο είναι οι νέες χώρες μέλη. Η Ελλάδα όμως επίσης είναι από τις χαμηλότερες χώρες χρησιμοποίησης των σχημάτων ΕΕΔ. Στα διαμεθοριακά ΕΕΔ τώρα κάναμε μία σειρά μελετών αναπερίπτωση καταρχήν 7 εθνικά προγράμματα ΕΕΔ διαμεθοριακά και τρία πανενουσιακά. Το EECCNet που είναι για τους καταναλωτές, το FinNet για τα δημοσιονομικές διαμάχες και το Solvit που είναι δίκτυο που επιλύει διαφορές που αφορούν την κακή εφαρμογή του, της ενωσιακής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν διαφορές βέβαια και ως προς τον αριθμό των περιπτώσεων η χαμηλότερη χρήση ήταν λίγο κάτω από τις 3.000 και η υψηλότερη το 2010 163.000. διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν και φραγμοί στη χρήση του ΕΕΔ. Για τις επικαλύψεις που υπάρχουν ανάλογα με το εθνικό ή το υπερεθνικό πρόγραμμα βρίσκουμε διαφορές και ανατομέα και αναπεριφέρεια. Δεν γνωρίζουν όλοι πάντοτε την ύπαρξη αυτών των διαδικασιών και πολλές φορές γι' αυτόν τον λόγο οι επιχειρήσεις διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν και άλλοι φραγμοί, η, ο γλωσσικός και η απουσία, η σωματική απουσία του καταναλωτή από τη χώρα όπου γίνεται η επιχείρηση. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα προγράμματα ε, ε, εδώ δεν δέχονται προσφυγές ή παράπονα από τρίτες χώρες. Αν κάποιο θέλει να υποβάλει παράπονο για επιχείρηση που δεν ε, εδρεύει στη χώρα του, δεν γίνεται δεκτό το παράπονο. Δεν υπάρχει δηλαδή αρκετή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, ούτε είναι κανείς βέβαιος ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί δεσμευτικά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εθελοντική νομολογία, όπως του διαμεσολαβητή, πολλές επιχειρήσεις εθελοντικά υποβάλλονται σε αυτές τις διαδικασίες και υπάρχει και το σουηδικό πρόγραμμα που παίρνει αποφάσεις αναπερίπτωση και τις αποφάσεις του τις βασίζει είναι και αυτές θελοντικές. τώρα για τα δίκτυα ενωσιακά δίκτυα το Solvit έχει διαφορετικό αντικείμενο αλλά δίνει και αυτό κάποια μαθήματα ιδιαίτερα από ότι είναι χρήσιμο ένα συγκεντρωτικό σύστημα ηλεκτρονικής δικτύωσης. Στο FinNet διαπιστώσαμε ότι θεωρείται χρήσιμο από όσους το χρησιμοποιούν και από τους καταναλωτές αλλά έχει πολλές ελλείψεις, δεν τα καλύπτει όλα γεωγραφικά. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι το ECC Net παίζει τον σημαντικότερο ρόλο διαμεθοριακά χρησιμοποιούν ένα συγκεντρωτικό και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης των παραπώνων γεφυρώνουν ε, τα γλωσσικά χάσματα και προβλήματα και παρεμβαίνουν άμεσα αν δεν υπάρχει άλλο σύστημα ΕΕΔ χορηγώντας πληροφορίες και βοήθεια. Το ECC στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκπαιρέωσε 800 περιπτώσεις το 2010, αλλά μόνο 24 από αυτές χρησιμοποιούσαν υπάρχοντα σχήματα ΕΕΔ. Τέλος, η χορήγηση πληροφοριών και βοηθείας για τις δυνατότητες επίλυσης διαφορών είναι σημαντικό στοιχείο του ECCNet. Για την νομική ανάλυση εξετάσαμε τρία σχήματα, το ECCP, την ε, οδηγία διαμεσολάβησης και την οδηγία για τα ασφαλιστικά μέτρα. Συγκρίναμε την, ε, τον τρόπο εφαρμογή της με από διάφορα κράτη και τη χρήση του από τους καταναλωτές. Η εφαρμογή λοιπόν σε πέντε χώρες μέλη, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, για το ESCP χρησιμοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η οδηγία Injunctions για τα ασφαλιστικά μέτρα έχει πλήρως μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των, αυτών των χωρών και η οδηγία για τη διαμεσολάβηση υποτίθεται ότι θα είχε μεταφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 21 Μαΐου 2011 αλλά στις άλλες χώρες μέλη δεν έχει ακόμα γίνει η μεταφορά ή δεν έχει ακόμη γίνει η τελική έγκριση. Κάθε φορά που εξετάζαμε τη χρήση, κάθε φορά που το ενωσιακό εργαλείο αφήνει κάποιο περιθώριο στα κράτη-μέλη, εκεί βλέπουμε να σημειώνονται σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το εργαλείο αυτό εθνικά. Η χρήση από τους καταναλωτές τώρα. Πρώτον, γενικότερα, έχουμε περιορισμένο αριθμό δεδομένων. Αυτό μας εξέπληξε γιατί δεν ήταν πάντοτε σαφής η πληροφόρηση που μας δόθηκε και κυρίως δεν ήταν συστηματική. Χαρακτηριστικά δεν, έγινε, δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση μεταξύ των αντικειμένων των παραπώνων και δεν μπορέσαμε άρα να ταυτίσουμε το είδος των προσφυγών. Καταλήξαμε λοιπόν ότι για το ESCP αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ λίγο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία το 2010 μόνο 36 αιτήσει υποβλήθηκαν, ενώ στην Ολλανδία το 2009 και 10 μόνο 10 και 20 αναλόγως. Οι λόγοι για αυτό τον περιορισμένη χρήση θα μπορούσαν να είναι πρώτον ότι δεν είναι γνωστή η ύπαρξη του εργαλείου αυτού και δεύτερον ότι μπορεί να έχει ελλείψει το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτές οι ελλείψεις λοιπόν τις ταυτίσαμε ως εξής. Πρώτον για το ESCP Πρώτο πρόβλημα. Δεν υπάρχει διαφάνεια για το κόστος της διαδικασίας. Όταν ένας καταναλωτής υποβάλλει προσφυγή που αφορά ας πούμε 2.000 ευρώ πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο θα είναι το κόστος. Πρέπει να είναι χαμηλό αλλά να υπάρχει και προβλεψιμότητά του. Δεύτερη έλλειψη, το έντυπο της Καμιά φορά πρέπει να συμπληρώνεται σε γλώσσα άλλη από, από τη μητρική του καταναλωτή. Και αυτό θέτει προβλήματα. Γιατί ορισμένα μέρη του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν από τον καταναλωτή και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει σε άλλη γλώσσα. Υπάρχει επίσης έλλειψη σαφήνειας και νομικής σαφήνειας ιδιαίτερα. Δεν είναι σαφές για τον καταναλωτή όχι μόνο για το ποιο θα είναι το κόστος της διαδικασίας αλλά και πόσο θα κρατήσει. Δεύτερον, η οδηγία για τη διαμεσολάβηση. Ποιες είναι οι δικές της ελλείψεις. Πρώτον, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει επικάλυψη, να εφαρμόζονται διαφορετικά συστήματα, ένα εθνικά και ένα διαμεθοριακά, άλλο διαμεθοριακά. Γιατί το βλέπουμε αυτό σαν πρόβλημα, διότι και αυτό καθιστά τα πράγματα ασαφή για τον καταναλωτή. Δεύτερον, δεν υπάρχουν υποχρεωτικά πρότυπα ως προς την ποιότητα των διαμεσολαβητών της διαμεσολάβησης και τρίτον υπάρχουν εκκρεμή προβλήματα πάλι το γλωσσικό ποιος θα πληρώσει τον διαμεσολαβητή και πόσο θα χρειαστεί να πληρώσει. Όσο για την οδηγία των ασφαλιστικών μέτρων, πρώτον διαπιστώσαμε ότι δεν έχει και πολλά δεν είναι και πολύ αποτελεσματική, δεν προβλέπει αποσημείωση δηλαδή και υπάρχουν πολλές διαδικαστικές διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Διαφορετικές κυρώσεις και μεγάλη ασάφεια ως προς το κόστος πάλι. Τέλος, και τα τρία αυτά εργαλεία έχουν ένα κοινό στοιχείο. προϋποθέτουν την ε, δικαστική προσφυγή. Δεν είναι δηλαδή πραγματικό σύστημα αποφυγής του δικαστηρίου. Απλώς συμπληρώνει τη δικαστική διαδικασία. Και τώρα ερχόμαστε στο τμήμα που αφορά τον Φρανκ. Αφού λοιπόν είδαμε ποιες είναι οι ελλείψεις και τι ισχύει, πρέπει να δούμε πρώτον τι μπορεί να γίνει. Πρώτον, δεν υπάρχει ειδικό νομικό εργαλείο στην Ένωση για να διευκολύνει τη διαμεσολάβηση σε διαμεθοριακά προβλήματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Σε μερικές χώρες ισχύει αυτορύθμιση και συνρύθμιση, αλλά αυτό είναι μάλλον εξαίρεση παρά ο κανόνας. Υπάρχοντες μηχανισμοί ΕΕΔ που βασίζονται σε αυτορύθμιση συνήθως δεν αφορούν όλους τους εμπορευόμενους. Ας πούμε το μικρεμπόριο δεν καλύπτεται. ή απαιτείται να είναι κανείς μέλος μιας επαγγελματικής οργάνωσης. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του. Σε ορισμένους μόνο τομείς υπάρχει μεγάλη πρόσβαση όπως στις τηλεπικοινωνίες όπου υπάρχει σαφές νομικό υπόβαθρο. δεν, έχει μιμηθεί, δεν έχουν μιμηθεί οι υπόλοιποι τομείς αυτούς όπου χρησιμοποιείται η τέτοια διαμεσολάβηση. Για τα χρηματοπιστωτικά ας πούμε δεν ισχύει ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης είναι ενδιαφέρον τομέας για τέτοια επίλυση διαφορών. Χρειάζεται λοιπόν κάποιο ειδικό νομικό εργαλείο ιδιαίτερο. Θα λέγαμε ναι. Και θεωρούμε ότι μεταξύ τομέων θα μπορούσε η επίλυση διαφορών να επεκταθεί. Θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση, η καλύτερη πρόσβαση σε διαμεθοριακά συστήματα τέτοιας επίλυσης διαφορών θα ήταν κάτι το ενδιαφέρον αν καλύπτουν, αν καλύπτουν τα συστήματα αυτά περισσότερες περιφέρειες και να μην περιορίζονται μόνο στα διαμεθοριακά θα μπορούσαν να γίνουν οικονομίες αν λυνόταν και τα προβλήματα της γλώσσας και αν υπάρχει κρίσιμη μάζα βέβαια που να διασφαλίζει στους καταναλωτές την πρόσβαση γιατί μπορεί να υπάρχουν αυτά τα συστήματα αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα ή για έναν μεμονωμένο τομέα και αυτό δεν ωφελεί τους καταναλωτές ούτε τις καταναλώτριες. Επίσης είναι σημαντικό αφού μιλάμε για νομοθετική δράση σε ενωσιακό επίπεδο θα έπρεπε να υπάρχουν πολλαπλές προσεγγίσεις Τα συστήματα που λειτουργούν καλά παρόλα αυτά, γι' αυτά οι καταναλωτές φοβούνται μήπως ζημιώσουν τελικά από τη χρήση τους λόγω της ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων μεταξύ χωρών μελών. Πρέπει λοιπόν να βασίζεται η αξιολόγηση όχι στις προβλεπόμενες διαδικασίες αλλά στο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν θα μπορούσαν όχι δεσμευτικά να βγάζουν αποφάσεις με συστάσεις, με συμβουλές, με κατευθυντήριες γραμμές και οι χώρες μέλη που δεν έχουν πλήρη συστήματα διαμεσολάβηση τέτοιας επίλυσης των διαφορών να μπορούν να επιλέξουν το πρότυπο που τους ταιριάζει περισσότερο. Αν δούμε τώρα ορισμένα παραδείγματα βελτίστων πρακτικών, πολλές φορές αναρωτιούνται οι καταναλωτές αν το πρόγραμμα, το, η διαδικασία προβλέπεται από υπάρχουσες οργανώσεις καταναλωτών, αν υπάρχει ή όχι ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης γιατί οι καταναλωτές θα ωφελούνταν από την ύπαρξη ενός τέτοιου ενιαίου single entry point όπου να μπορούν να απευθυνθούν για να υποβάλουν παράπονα ή και απλώς για να πληροφορηθούν διότι η κύρια λειτουργία ενός τέτοιου ενιαίου σημείου πρόσβασης θα ήταν να οδηγήσει τον καταναλωτή που να αποφθυνθεί. Η πρώτη επαφή είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου και έπειτα η συλλογή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών θα ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για να δούμε πώς χειρίζονται τα παράπονα και τις προσφυγές των καταναλωτών. Τώρα η πρόσβαση σε ΕΕΔ, σε διαμεθοριακά θέματα και πάλι το ενιαίο σημείο πρόσβασης θα ωφελούσε τον καταναλωτή και είναι πολύ πιθανό ένα τέτοιο μελλοντικό ενιαίο σημείο πρόσβασης να βοηθήσει ιδιαίτερα για τη συλλογή στοιχείων και για τη δημιουργία επαφών μεταξύ χωρών μελών, μεταξύ εμπορευομένων για να μπορέσουν να επιλύσουν μια διαφορά πιο αποτελεσματικά. Γιατί πριν γίνει το πράγμα επίσημο υπάρχει πάντοτε μια ανεπίσημη πρώτη φάση πληροφόρησης. Πρόσβαση λοιπόν και σε μηχανισμούς ε, ε, εδώ σε άλλες χώρες μέλη. Πράγμα το οποίο παρεμποδίζεται αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει ούτε γνώση για την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων, υπάρχει και ο γλωσσικός φραγμός. Θα μπορούσε να, υπάρχει, να δημιουργηθεί ένα πρότυπο έντυπο που να χρησιμοποιείται παντού. Ας πούμε τα αγγλικά να χρησιμοποιούνται για όλα τα έντυπα σε διαμεθοριακές διαφορές ή ηλεκτρονικά ή μη ηλεκτρονικά. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η γνώση της ύπαρξης των συστημάτων αυτών. Επειδή όμως υπάρχει κατακαιρματισμός και ελλείψη στην κάλυψη στον αριθμό χωρών που εφαρμόζουν τέτοια συστήματα, θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι το να προωθήσουμε απλώς την ύπαρξη των συστημάτων να τα διαφημίσουμε δεν αρκεί. Πρέπει πρώτα να βελτιωθούν οι υποδομές, τα ίδια τα προγράμματα και οι διαδικασίες σε κάθε χώρα μέλος. Οι χώρες που έχουν ένα ενοποιημένο σύστημα επίλυσης διαφορών, εναλλακτικών επίλυσης διαφορών, είναι λίγες όταν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα το γνωρίζουν και οι καταναλωτές σχεδόν αυτόματα. Το, δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτό το πρώτο βήμα τέλος. Κάτι που δεν πρέπει επίσης να ξεχάσουμε είναι το θέμα των πόρων που πρέπει να δώσουμε σε αυτά τα συστήματα. Ορισμένα χρειάστηκε να λήξουν γιατί δεν είχαν πόρους στη διάθεσή τους. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν βιώσιμη χρηματοδότηση για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ιδιαίτερα σε διαμεθοριακά προβλήματα όπου το κόστος είναι υψηλότερο λόγω των μεταφράσεων. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη είτε μέσω άμεσης δημόσιας χρηματοδότησης είτε μέσω κάποιας φορολόγησης των επιχειρήσεων ή εισφοράς ή μέσω των αποζημιώσεων που θα δίνονται ως αποφάσεις δηλαδή στο επίπεδο της επιχείρησης. Πολλές επιχειρήσεις με χαρά θα δέχονταν να χρηματοδοτήσουν ένα τμήμα τέτοιων διαδικασιών προκειμένου να επιληθούν οι διαφορές εκτός δικαστηρίων. Τέλος, η ανεξαρτησία της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να παρεμποδίσει να, τη, χρηματοδότηση, δεν πρέπει η χρηματοδότηση μάλλον να παρεμποδίσει την ανεξαρτησία των διαδικασιών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Έχω ένα δίλημα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Θέλω να ρωτήσω ε, τον εισηγητή. Ε, ο κ. Ροσφόρ είναι εδώ. Ε, ίσως θα θέλατε κ. Σιγητά να απαντήσετε σε ορισμένα από τα πορίσματα της μελέτης και να, αναφέρετε, να μας παρουσιάσετε και τη δική σας έκθεση. Και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις για να σχολιάσουν και τα δύο πράγματα. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε ε, να ζητήσουμε και απαντήσεις από, τις, από την ομάδα των μελετητών. Ε, δεν έχουμε και πολλά, πολύ χρόνο βέβαια, συμφωνείτε όμως με αυτή τη διαδικασία. Να δούμε παράλληλα και την έκθεση και τη μελέτη. Ωραία. Ο κ. Ροσφόρ θα μιλήσει πρώτος. Ο κ. Φόξ είναι εδώ, ο κ. Τριανταφυλλίδη είναι εδώ. Να δούμε το εκπροσώπηση και των άλλων ομάδων ενδεχομένω. Ο κ. Μπιτμάγερ. Δεν ξέρω αν κάποιο από το ΕΛΚ θέλει να πάρει το λόγο. Ο κ. Ζουρά είναι εδώ. Θα δούμε. Ο κ. Ροσφόρ έχει καταρχήν το λόγο. Έχετε δίκιο. Για λόγους ταχύτητος ε, θα κάνω την έκθεση της έκθεσής μου και μέσα στα σχόλιά μου θα κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις για την μελέτη που μας παρουσιάστηκε. Καταρχήν να πω ότι η μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά χρήσιμη επιπλέον. Ε, σπάνιο φαινόμενο. Λοιπόν, το ποιο είναι το πλαίσιο. Πρόκειται για μια έκθεση γνωμοδότησης για τις, ε, τα συστήματα επίλυσης διαφορών προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, έχει, βλέπει το θέμα με ένα πιο, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Καταρχήν εισαγωγικά. Κάτι που έχει σχέση και με τη μελέτη που μας παρουσιάστηκε. Βλέπουμε ότι τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών λειτουργούν και λειτουργούν όλο και περισσότερο. Και η μελέτη επιβεβαιώνει ότι αυτό που προτείνω και εγώ, ε, βέβαια ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την επιθυμία της Κομισιόν να ενθαρρύνουμε τα συστήματα αυτά, να λειτουργήσουν καλύτερα με νομοθετικές προτάσεις πριν το τέλος του έτους και να τα θεωρήσουμε, όπως τα έχει θεωρήσει και η Κομισιόν, ως προτεραιότητα για την ε, Single Market Act που συζητείται αυτή τη στιγμή. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Η μελέτη το απέδειξε και εμείς επίσης το επιβεβαιώνουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και από πλευρά τομέων και από γεωγραφικής πλευράς. Οπότε θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε για την προώθηση του συστήματος. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ε, χρησιμοποίηση του συστήματος μεταξύ των χωρών που έχουν χαμηλούς δείκτες είναι και η δική μου χώρα. Και αυτό αποδεικνύει ότι θα πρέπει να καλύψουμε καλύτερα τομεακά και γεωγραφικά ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ας δούμε την ουσία του θέματος. Η μελέτη κατέδειξε την ε, μεγάλη ποικιλία υποθέσεων από τα, είδαμε τα 750 παραδείγματα και είναι ενδιαφέρον που η μελέτη ε, λέει πως δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες για όλες αυτές τις υποθέσεις συνεπώς χρειαζόμαστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία Πράγματι, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή, ενιαία ευρωπαϊκή χάρτα πάνω στην οποία να βασίζονται τα συστήματα εναλλακτική επιλύση διαφορών. Αυτό δεν σημαίνει κανονισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε τα ίδια συστήματα, απλά θα πρέπει να οργανώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ιδέες που διέπουν τα ε, συστήματα ε, εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Και ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα, πρέπει να είναι τα κεφάλαια αυτής της χάρτας. Τρεις κατηγορίες κεφάλαιων. Πρώτη κατηγορία, τα, ε, τα απλουστευμένα συστήματα τα απλά συστήματα. Ε, καταρχήν, τα ΕΕΔ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και γρήγορα. Συνεπώς, αυτή, ε, αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα και τις αρετές, ίσως το πιο βασικό πλεονέκτημα των συστημάτων. Ε, Συνήθω λέμε ότι οι διαδικασίε αυτές είναι διαδικασίε ισότιμε. και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αν δεν εξασφαλίσουμε την, ισότιμ, την ισοτιμία, ε, την ε, ε, ισορροπία θα καταρρεύσουν. Αν ο κόσμος αντιληφθεί ότι δεν είναι δίκαια και ισότιμα δεν θα καταφέρει σε αυτά. Ε, μετά, ο σεβασμός ε, της καταδικής τη απόφαση, κοινό σε όλα τα συστήματα, η ελευθερία και ο θελοντικός χαρακτήρας τους. Επειδή πρόκειται για εξοδικαστική ρύθμιση διαφορών, δεν ε, ε, είναι αντιφατικό να θέλουμε να επεκτείνουμε τα συστήματα αυτά γεωγραφικά και τομεακά και ταυτόχρονα να, τα διατηρήσουμε, ε, να διατηρήσουμε τον εθελοντικό τους χαρακτήρα. Όλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα παρόλα αυτά να καταφύγουν, να προσφύγουν συγγνώμη, σε ένα δικαστήριο. Τέλος, ε, παρόλο που η ομάδα μου είναι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το θέμα, επιμένω στην αναλογία των αποφάσεων και του κόστου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι πολύ σημαντικό να το καταγράψουμε και ω κοινό παρανομαστή των αναλυτικών ε, συστημάτων επίλυσης διαφορών. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μας βρουν σύμφωνους. Δεύτερο τμήμα πληροφοριών που θα πρέπει να καταγράψουμε είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην ίδια την έκθεση προτείνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ε, εναλλακτικέ λύσεις για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Ενδεχομένως δεν θα μας βρουν όλους ε, σύμφωνους, αλλά που θα μπορούσαμε να τις ε, συμφωνήσουμε τελικά, γιατί κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικές. Τι εννοώ. Πρώτον, το θέμα της διαφάνειας και της ανάγκης ετήσιας έκδοσης εκθέσεων. Το λέτε και εσείς στις προτάσεις σας στη μελέτη. Ίσως ήμουνα ε, ιδιαίτερα συντηρητικό στην εκθέσή μου. Εγώ δεν λέω ότι χρειάζονται αιτήσει εκθέσει, ούτε και αναφέρω στην έκθεσή μου ε, ποια θα πρέπει να είναι η μορφή του. Εσεί στη μελέτη σα καταδεικνύονται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ. Ε, υπάρχουν περιπτώσει που τα συστήματα επίλυση διαφορών δείχνουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ΟΜΑ ε, και άλλες περιπτώσεις που δεν ε, λαμβάνει η χώρα μια τέτοιου είδους ε, πράξη, αλλά θα χρειαστούμε αυτές τις εκθέσεις. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει τα συστήματα να είναι δωρεάν, όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο αριθμό των περιπτώσεων ήδη. Όλοι άλλωστε οι ενδιαφερόμενοι, ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, και οι οργανώσεις καταναλωτών ε, είναι υπέρ του ε, δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερο τρόπο οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα συστήματα και να τα εμπιστεύονται. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα μικρό αποτρεπτικό κόστος. Τρίτη σειρά σημείων Ε, για τα οποία χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο. Τα συμπεριέλαβα στην έκθεσή μου και περιμένω να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων, των σχεδόν εισηγητών και των μελών της Επιτροπής μας. Πρώτον, η ποικιλομορφία και η ποικιλία των διαμεσολαβητών. Πιστεύω ότι οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να προέρχονται από τον ε, τομέα των επιχειρήσεων αλλά και από τον τομέα των καταναλωτών. Και για αυτά τα για να αντιπροσωπεύει κανείς όλα αυτά τα συμφέροντα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα. Θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι ικανοί και γι' αυτό λόγο κάνω δύο προτάσεις. Πρώτον, να δίδεται μια κατάρτιση στους διαμεσολαβητές. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα για τις αγωγές των ε, καταναλωτών που ε, συγγνώμη, ιδιαίτερα για, τις, ε, για τους καταναλωτές ε, που θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Επίσης χρειάζεται να δίδεται και μια πιστοποίηση ISO. ISO. Μετά, πολλές φορές κάνουμε λόγο για την αμεροληψία των ε, διαμεσολαβητών. Εσείς μιλάτε στην έκθεσή σας για την ανεξαρτησία τους. Και η κυρία Ουάλης χρησιμοποιεί στην έκθεσή της την ίδια έκφραση. Πέραν όμως ε, του, του, τύπου, η ανεξαρτησία είναι πιο ισχυρή έννοια από την αμεροληψία. Δηλαδή η ανεξαρτησία ε, υποδεικνύει μια μεγαλύτερη απόσταση από τα συμφέροντα τα οποία κρίνει ο διαμεσολαβητής. Ε, υπάρχει και το θέμα των διαμεσοριακών ε, διαφορών. Ξέρετε, το λέτε και εσείς ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο. Χρειάζεται ένας πρόσθετος μηχανισμός. Ε, δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Είναι πιο περίπλοκο. Ίσως θα έπρεπε τα κλασικά συστήματα επίλυσης διαφορών να μην επιλαμβάνονται ε, τέτοιου είδου ε, διαφορών ε, τα οι οποίες θα μπορούσαν να ρυθμιστούν μέσω μιας ενιαίας στηρίδας κλπ. νομίζω ότι τα συστήματα των τα αναλυτικά συστήματα επίση διαφορών είναι κατάλληλα, λειτουργούν και τέλος ένα τελευταίο σχόλιο και προς την Κομισιόν μια πρόταση για την ακρίβεια ίσως θα έπρεπε να δούμε την, τον όρο όταν ο όρος αυτός μεταφράζεται στα γαλλικά ή σε άλλες γλώσσες από τα αγγλικά, ε, μεταφράζεται αρνητικά. Ε, ο καταναλωτής ε, δεν καταλαβαίνει τι είναι, σε τι είναι εναλλακτικά αυτά τα αισθήματα, εναλλακτικά είναι τίνος. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για φιλική επίλυση διαφορών ή διαμεσολάβηση επίλυσης διαφορών έτσι ώστε οι κατανοητέ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ. Σα uh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ περιεκτική η απάντησή σας. Ε, διάβασα καλά ε, το έγγραφο που μας έχετε καταθέσει ε, και σήμειωσα κυρίως αυτά που είπατε για το χάρτη πραγματικά εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο κύριος Άλεβα, δηλαδή ότι τα νομοθετικά εργαλεία θα πρέπει να εστιάζονται περισσότερο στο αποτέλεσμα και όχι τόσο στη διαδικασία. Και νομίζω αυτό είναι και το οδηγό νήμα που διατρέχει τη δική σας την ε, τοποθέτηση. Κύριε Μάιερ, δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε πρώτο το λόγο, ε, γιατί δεν ήσασταν εδώ, ίσως να μην ακούσατε το μεγάλο μέρος των προσεγγίσεων. Η κύριε Βάιλερ και μετά ο κύριος Μάιερ και μετά ο κύριος Φόξ και κατόπιν ε, θα δούμε ε, πώς θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κυρία Βάιλα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν, δεν δίστανται κατά πολύ οι απόψει ε, της δικής μου της πολιτικής ομάδας από αυτές του εισηγητή. Έχουμε όμως κάποιες ερωτήσεις. Η πύληση διαφορών, η εκεί όπου έχει εισαχθεί, όπου είναι γνωστή και όπου λειτουργεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Είναι ευέλικτη, ταχύτατη, προσιτή στο κόστος, όχι απαραίτητα ε, γνωστή σε όλους, αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί και για τους καταναλωτές και για την οικονομία. Και έχω λοιπόν την εξής πρώτη ερώτηση. Έχετε κάνει εμπειρία και με public to business. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία έχουμε μία σειρά διαδικασιών, ε, διαιτησιών ε, ανάμεσα σε κράτος ε, και εργολάβους, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όπου η διαιτησία είναι λιγάκι διαφορετική, όχι ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πελάτες, καταναλωτές, αλλά στο δημόσιο και επιχειρήσεις. τώρα, κάτι άλλο που δεν το κατάλαβα καλά. Χρειαζόμαστε πράγματι νομοθετική πρόταση ε, πολλοί με τους οποίους ε, συζήτησα μου είπαν ότι οι προτάσεις πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αρκούσαν και δεν χρειάζεται απαραίτητα νομοθετική πρόταση. Εγώ όμως είμαι ανοιχτή, δηλαδή αν ε, η Νομική Επιτροπή και η δική μας Επιτροπή καταλήξουν στο ότι πράγματι χρειαζόμαστε νομοθετική πρόταση, γιατί όχι. Συμφωνώ όμως και με τη δική σας άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο, δηλαδή να υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία χωρίς να υπάρχει τίποτα ε, τίποτα απολύτω όπως στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και ίσω και επικίνδυνο. Και άλλη ερώτηση. Η Τράπεζα Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκεί. Δεν μπόρεσα να τη δω, αλλά αυτό που θα βοηθούσε εμά είναι να υπάρχουν οι βέλτιστες ε, πρακτικές ε, από ορισμένα κράτη-μέλη, κυρίως σε online συνδέσεις, κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Η επόμενη ερώτηση αφορά τον εισηγητή. Ε, στην εισαγωγική σας παρατήρηση αναφέρεστε σε μια νομοθετική πρόταση και παράλληλα λέτε να υπάρχει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χάρτης. Αυτό όμως για μένα είναι αντίφαση. Ενιαίος ευρωπαϊκός χάρτης, αυτό έτσι πολύ μεγάλη επίβολα, αλλά αν τελικά το έχουμε αυτό ή για να το πω αλλιώς λέει ο Μιλήτρια, ή ο χάρτης δεν περιέχει τη νομοθετική πρόταση. Δεν καταλαβαίνω καλά τι ακριβώς λέτε με αυτό το χάρτη. Αναφέρεστε σε ανεξαρτησία. Και όσον αφορά την ε, τεχνογνωσία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Προφανώς και χρειαζόμαστε προδιαγραφές και οικονομική ανεξαρτησία η οικονομική απαλλαγή για τους καταναλωτές συμφωνώ απόλυτα μαζί σας μόνο που είπατε στην παρέμβασή ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν κοιτάξτε δεν είναι δυνατόν να είναι όλα δωρεάν ε, πρέπει να πούμε να είναι δωρεάν για τον καταναλωτή και στις ε, οικονομικές ενώσεις υπάρχει ε, μια ε, εισφορά αλληλεγγύης του κλάδου που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους διαδικασίες δεν νομίζω ότι σε κράτη που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το κόστος να μετακυλιστεί στο κράτος. Όχι δηλαδή να πληρώνει ας πούμε, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, να πληρώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη που ενδιαφέρονται με αυτόν τον ταχύτατο τρόπο να διευθετηθεί η διαφορά τους. Και ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη, αυτή είναι η οικονομική κύκλη. Εντάξει, δωρεάν για τον καταναλωτή, αλλά και κάποιο πρέπει να πληρώνει το προαιρετικό στοιχείο. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και η δυνατότητα σε ε, διάφορα στάδια της ε, διαδικασίας ε, να μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η φιλική αυτή διευθέτηση. Τώρα δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε στα δικαστήρια αναφερθήκατε σε αυτή τη σφραγίδα ποιότητας την ευρωπαϊκή. Για μένα αυτό είναι ένα κριτήριο ποιότητας, όπως και ο χάρτης. Ίσως λιγάκι πρέπει να το προβλέψουμε αυτό. Ε, τελειώνω σιγά σιγά. Στη Γερμανία έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα δημόσιου και ιδιωτικού δημόσιων και ιδιωτικών αρμόδιων αρχών. Στη Γερμανία αυτό το σύστημα έχει αποδειχθεί πάρα πολύ καλό και δεν θέλουμε να το ε, αλλάξουμε. Εμείς στη Γερμανία βελτιώσαμε και το σύστημα των διαμεσολαβητών. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν θέλουμε να υπάρχει ένας και μόνο φορέας. Για τις διασυνοριακές διαφορές, εκεί εντάξει να υπάρχει ένας φορέας. Όμως σε τοπικό επίπεδο όπου οι ε, ε διαφορές διευθετούν ταχύτατα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διάφοροι, περισσότεροι από έναν αρμόδιοι φορείς. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του έτους και ίσως ε, είναι δυνατόν την ομιλία σας ε, να τη μεταφράσουμε σε περισσότερες γλώσσες γιατί όχι και το σύνολο της μελέτης και αν όχι το σύνολο της μελέτης τότε ε, την περίληψη, τα συμπεράσματα της μελέτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, αναγκάστηκα να πάω ε, σε μια πολύ σημαντική συζήτηση και να φύγω από την αίθουσα, αλλά είχα αφήσει τη συνεργάτη μου και θα με ενημερώσει. Ε, κάποιες, ε, κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις. Συνάδελφε Ροσφόρ, πάρα πολύ καλή η έκθεσή σας, το σχέδιο της έκθεσης ε, και πολύ καλές και απόψεις που εκφράσατε, που και εγώ τις στηρίζω, όπως και η προλαλή σας. Να πω όμως και κάτι το να γνωρίζει κανείς τέτοιου είδους διαδικασίες, αυτό είναι το σημαντικότερο. Ε, το να αποφασίζουμε πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται, τι νόημα έχει αυτό. Και βλέπουμε αυτό ε, συμβαίνει και στη Γερμανία, αυτή η διευθέτηση μικρών διαφορών. Ε, ούτε καν τα δικαστήρια δεν το γνωρίζουν αυτό, ούτε υπάρχουν έγγραφα, μηχανία, χάος. Επίσης, όσον αφορά τις εξαιρετήσεις ενημέρωσης, συμφωνώ. Η Τράπεζα Δεδομένων της Επιτροπής ε, είναι πολύ περίπλοκη. Έχουμε εδώ να κάνουμε με καταναλωτές, δεν έχουμε να κάνουμε με νέους ε, που είναι εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε λίγες ιστοσελίδες, αλλά σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εύκολα link. Πρέπει επίσης ε, να είναι όλα αυτά προσαρμοσμένα στον πολύ απλό καταναλωτή, κατά πόσο μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, πώ μπορούμε να τον ενημερώσουμε, πού βρίσκεται, σε ποιες γλώσσες. Δεύτερη παρατηρήσή μου. Νομίζω ότι ορισμένες έννοιες πρέπει να τις συγκεκριμενοποιήσουμε. Βεβαίω, εγώ ως νομικός ενδιαφέρομαι στο να, για το να, έχω, να έχουμε τις ε, ε, σαφέστερες δυνατές ε, διευκρινήσει, ορισμού που να μπορούν να του ε, χρησιμοποιήσουν οι δικαστέ. Παραδείγματο χάρη, τι σημαίνει επαγγελματική οργάνωση. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε. Ε, περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνει τις μικρομεσαίες. Μήπως πρέπει να προβούμε σε κάποια διαφοροποίηση. Επόμενη παρατήρησή μου αφορά σε κάτι ε, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Ανεξαρτησία, αμεροληψία, αρμοδιότητα. Όμως για να αποκτήσει κανείς ε, αρμοδιότητα εμείς ε, θέλουμε να έχουμε ω δυνατόν περισσότερους διαιτητές. Όχι ένα για τη Γερμανία Γερμανία και ένα για τη Γαλλία, αυτό όμω κοστίζει και ποιο θα το πληρώσει. Και αν δεν το πληρώνει το κράτο, πρέπει να το πληρώνουν οι επιχειρήσει. Άλλη ερώτηση. Μα ποια επιχείρηση, μια επιχείρηση με δύο άτομα, αυτή δεν μπορεί να πληρώσει. Και παρόλα αυτά όμω μπορεί να προκύψουν και σε αυτή την επιχείρηση των ε, δύο τόμων ε, να προκύψει κάποια διαφορά για τα προϊόντα τη. Άρα δηλαδή να συνδυάσουμε τον ορισμό με την αρμοδιότητα και το κόστο. Αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε. Όσον αφορά τώρα ε, το δωρεάν τη όλη διαδικασία. υπάρχει κίνδυνο, κοιτάξτε αν κάτι είναι τελείω δωρεάν είτε δεν αξίζει τίποτα ή ε, δεν το χρησιμοποιεί κανεί. αυτό έτσι είναι, είναι ανθρώπινο το ερώτημα κατά πόση ε, πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι 20 ή 50 ευρώ ε, που θα επιστρέφονται όπως και στις δικαστικές διαδικασίες της δίκης δηλαδή αυτό ισχύει μια τέτοια διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ ακριβή, γιατί ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει ή έστω και διαμεσαλαβητής να χρησιμοποιήσει ένα εμπειρογνώμονα που μόνο αυτός είναι αρμόδιος για να επιλύσει μια διαφορά. Η αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη είναι όποιος κερδίζει τη νίκη απαλλάσσεται από δαπάνες και όποιος χάνει τη δίκη καλύπτει το κόστος. Αυτό είναι σαφές. Αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι τελικά θα πλέον επιχειρήσεις ανεξάρτητα με το τι κοστίζει, πόσο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις ή πόσο δύσκολη είναι η υπόθεση. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε και να προβούμε σε μια διαφοροποίηση. Γιατί τελικά ε, δεν είναι σωστό ένας μικρομεσαίος ε, να καταθέσει, να ξεκινήσει μια ε, τέτοια διαδικασία αν όμως τελικά δεν κερδίσει τη νίκη να πρέπει να καλύψει το σύνολο των δαπανών. Δεν αυτό. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο και πραγματικά περιμένω να δω πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση. Γιατί πιστεύω ότι εδώ έχουμε κάτι το καλό που όλοι το επιθυμούμε και κατόπιν τούτου με αυτή την έννοια ενθαρρύνω τον εισηγητή να συνεχίσει περαιτέρω τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε μια σειρά ομιλητών στον κατάλογο κύριος Φόξ είναι ο επόμενος, ε, είναι η σκιώδη συγητής. Μετά έχουμε το, την κυρία Στάιλερ και τον κύριο Ζουβά. Ελπίζω ότι θα είναι σύντομη, γιατί έχουμε και άλλα δύο θέματα στην ημερησία διάταξη. Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης νομίζω. Α, μετά τον κύριο Φόξ θα είναι ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ε, και μετά η συγγένεια τη επόμενη ε, ε είναι. Ε, που είναι ίδια με αυτήν όσο λιγότερο χρόνο φάει τόσο περισσότερο θα έχει στην επόμενη έκθεση ευχαριστώ πολύ για τον, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ροσφόρ ε, Νομίζω ότι η προσέγγιση του για τη χάρτα είναι πολύ σωστή. Μίλησε για ένα σύστημα αποτελεσματικό, ρεαλιστικό, γρήγορο ε, και θελοντικής φύσεως. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, σε ό,τι είπε ο κύριος Μέιρ για το κόστος, να πω το εξή. Ίσως ε, υπερεκτιμάται, υπερβάλλεται σε ό,τι αφορά τα προβλήματα. Ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί ε, θα ε, ωφελεί τις επιχειρήσεις. Και αν δεν είναι δωρεάν δεν θα το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Το έχουμε δει αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν νομίζω ότι το σύστημα θα κατακλειστεί από ε, ψευδοαγωγές ε, και ψευδοπροσφυγές. Ε, ε, άλλωστε, αν έχουμε πολλές προσφυγές, αυτό θα σημαίνει ότι θα απελευθερωθούν πολύ τα δικαστήριά μας. Αν βάλουμε λοιπόν ένα αποτρεπτικό κόστος για την αρχή για την εκκίνηση μιας διαδικασίας, αυτό θα παρεμποδίσει πολλούς καταναλωτές και δεν θα το χρησιμοποιούν. Διαφωνώ με τον κύριο Ροσφόρο όμως σε ό,τι αφορά την παράγραφο 3 της νομοδότησής του. που λέει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογικών αγωγών είναι απολύτως απαραίτητο. Γνωρίζετε την ε, διαφορά μου, την ε, διαφωνία μου ε, θα το δούμε αργότερα, αλλά θα ήθελα να πω στη γραμματεία, μήπως θα μπορούσε να δει την αγγλική μετάφραση της παράγραφου 3, διότι είναι πραγματικά πολύ κακή. Το γαλλικό κείμενο είναι καλύτερο, αλλά το αγγλικό είναι απαράδεκτο. Ε, ακόμα και αν διαβάσετε από μόνοι σας την ε, παράγραφη της στα αγγλικά, δεν θα καταλάβετε το νόημά της. Λοιπόν, ας το κοιτάξει η γραμματεία παρακαλώ. Συμφωνώ με τον κύριο Ροσφόρ ότι τα εθνικά συστήματα θα πρέπει να, να συντονίζονται όταν εξετάζουν διαμεθοριακές διαφορές, αλλά ας αποφύγουμε τη δημιουργία ενός ακόμα ευρωπαϊκού οργάνου για την επίβλεψη του συστήματος. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ως λύση ε, μια ιστοσελίδα διαθέσιμη σε όλες τις, χώρες Ευρωπαϊκής, ε, σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ας αποφύγουμε λοιπόν την ε, περιττή γραφειοκρατία. Τώρα, η δημοσιοποίηση του συστήματος επίσης θα πρέπει να είναι αναλογική. Βέβαια, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα, αλλά δεν θα πρέπει να ε, υποβάλουμε σε υπερβολικό φόρτο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αυξήσουμε το κόστος για αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ροσφόρ. Πολύ καλή δουλειά του. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ. Ε, η παρουσίαση δεν ήταν τη Κομισιόν, ήταν των δικών μας των δικών μα συμβούλων. Ε, μάλλον κάνατε κάποιο λάθο. Εμεί τους πληρώσαμε. Ε, ο κ. Τρενταφυλλίδη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τους μελετήτε για την παρουσίαση της μελέτη, αλλά και τον συνάδελφο τον Ροσφόρ για την παρουσίαση τη έκθεση του και εμείς πιστεύουμε ότι οι μηχανισμοί εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προστασία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές βέβαια βρίσκουν σημαντικές δυσκολίες από τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένα πρότυπο για τα συστήματα εναλλακτική επίλυσης διαφορών. Αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να προωθούνται περισσότερο αφού σήμερα οι έμποροι δεν χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου μηχανισμούς και επιπλέον δεν έχουν κίνητρα να το πράξουν. Ω εκ τούτου η βελτίωση των μηχανισμών πρέπει να διασφαλιστεί αλλά και η σύνδεση του με του μηχανισμού συλλογική έννομη προστασία. Άλλωστε οι καταναλωτέ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύσουν τι διαφορέ του με τι επιχειρήσει με χαμηλό κόστο. Αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και θα τονώσει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίε που διεξάγονται εξ αποστάσεω ή και διαδικτυακά σημαντικά και να εξακολουθούν να υπάρχουν στα περισσότερα κράτη-μέλη, τόσο στην εφαρμογή όσο και στην πρόσβαση και επίσης επικρατεί η αντίληψη των καταναλωτών ότι σε μεγάλο βαθμό δεν φέρουν αποτελέσματα. Οι πιο πάνω προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο της Κομισιόν στην προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Um, uh, Ωραία. Κυρία Στάιλερ, ο κύριο Ζουβέν, κυρία Ράπτη, παρακαλώ εν συντομία. Και μετά θα επανέλθουμε στον εισηγητή. Ε, κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ στους συγγραφείς της ε, μελέτης και στους σκιώδης ηγητές. Κοιτάζοντας τις ε, διάφορες ε, χώρες, ε, βλέπετε ότι κάποιες χώρες έχουν 0 και κάποιες χώρες όπως η Γερμανία έχουν 233 υποθέσεις. Και εξετάζοντας τις τα στατιστικά για μικρές και μεγάλες ε, υποθέσεις βλέπουν ότι έχουμε διαφορές διότι δεν έχουμε τα στοιχεία από όλε τις χώρες. Είναι λίγο δύσκολο να συγκρίνουμε λοιπόν τα διάφορα συστήματα μεταξύ τους. Ε, είναι διαφορετικά και τα δικαιοδοτικά συστήματα. Συνεπώς να ρωτήσω το εξή. Ποια είναι τα τρία βασικά, ποιοι τρεις βασικοί, βασικοί τομείς ε, που καλύπτονται στην πράξη από τις αγορές από τις, ε, ε, από τις αγωγές. για παράδειγμα το, του, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου που σχετίζεται με τις διασυνοριακές επιλύσεις διαφορών είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Επίσης και ο κύριος Μάιερ μίλησε για το κόστος και άλλοι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι ανεξαρτήτως της απόφασης που θα πάρουμε για το κόστος δεν θα πρέπει το σύστημα να είναι εις βάρος της προσφυγής όλων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στο σύστημα. Ε... Ζουβάν. η φιλική επίλυση διαφορών νομίζω ότι ωφελεί όλους και την δικαιοσύνη ε, και τους ενδιαφερόμενους που επιλύονται διαφορές πιο γρήγορα και πιο οικονομικά ε, και βέβαια αποφεύγουμε ε, να έχουμε νικητές και ετημένους. Συνεπώς όλοι συμφωνούμε με τη φιλοσοφία. Τέσσερις ερωτήσεις, πέντε ερωτήσεις θέλω να θέσω στον κύριο Σφόρ. Πρώτον, ε, ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τη σύνδεση της παράφου 1 με την παράφου 6. Ή ζητούμε μια νομοθετική πρόταση ή ε, προχωράμε στην δημιουργία μιας χάρτας. Δεν καταλαβαίνω τις δύο αυτές προτάσεις παράλληλα. Δεύτερον, ε, το θέμα της πιστοποίησης ποιότητας. Ε, ποιος θα το κάνει αυτό, πώς θα ενοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία γνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων. Τρίτον, τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις φιλικές τα συστήματα φιλικής επίλυσης διαφορών και στις συλλογικές αγωγές. Ίσως θα έπρεπε να επιμείνουμε στο ότι οι συλλογικές αγωγές θα πρέπει να είναι η τελευταία εναλλακτική λύση αφού έχει εξαντληθεί η οδός της φιλικής επίλυσης διαφορών. Θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν στη χρήση τη διατησίας, της διαμεσολάβησης και μόνο να αποτύχει αυτή η λύση να έχουμε το θέμα των συλλογικών ε, αγωγών. Ε, επόμενο σχόλιο. Οι επιχειρήσει θα πρέπει να λάβουν τι ευθύνε του και να ενημερώνουν τον καταναλωτή για την ύπαρξη τέτοιων συστημάτων φιλική επίλυση διαφορών. Ε, να μην αφήσουμε το θέμα αυτό δηλαδή στα επιμελητήρια ή στι κρατικέ αρχέ μόνο. Ε, τέλος, συμφωνώ με τον δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος. αυτό θα επέτρεπε στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν περισσότερο το σύστημα. Mrs. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί νόμιζα ότι οι δύο εκθέσεις συζητούνται μαζί. Ε, εάν είμαι η τελευταία, ε, μπορώ να μην μιλήσω τώρα και να μιλήσω μετά με την έκθεσή μου. ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερο ό,τι διευκολύνει τη διαδικασία. Κοιτάξτε, θα έχουμε ξεχωριστή συζήτηση για τη δική σας την έκθεση. Τώρα συζητάμε για την έρευνα των μελετητών και την έκθεση του κυρίου Ροσφόρ. Ε, και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε σχόλια επ' αυτού. Συνεχίζω. Yeah. Ξέρετε, είχα στο μυαλό μου... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Μισό λεπτό. Λέμε ότι ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών και οι συλλογικές προσφυγέ πηγαίνουν χέρι-χέρι. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα ότι μπορεί να μιλάμε μαζί και ταυτοχρόνως για τις δύο εκθέσεις. Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι πολύ καλό αυτό που λέτε και συμφωνώ ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τα δύο θέματα. έρχομαι από, από μια ακρόαση που γίνεται με πρωτοβουλία της επιτροπής νομικών θεμάτων σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές και πρέπει να σας πω ότι και εκεί ε, οι συλλογικές προσφυγές με το ADR μπλέκονται με κάποιο τρόπο. Αυτό που ακούστηκε να λέει προηγουμένως ο κύριος Ζουβέν ως προβληματισμό μέχρι πού θα πηγαίνει το ADR και από πού και μετά θα πηγαίνουμε στις συλλογικές προσφυγές είναι κάτι που ε, συζητήθηκε αρκετά και σε αυτήν την ακρόαση. Ε, νομίζω ότι το δωρεάν στον εναλλακτικό μηχανισμό ε, βοηθάει. Βέβαια, έχω στο μυαλό μου και αυτό που είπε ο κύριος Μάγερ, ότι ό,τι δίνεις στο λαό δωρεάν έχει την τάση να το βλέπει με λιγότερη αξία από αυτήν που πραγματικά έχει ωστόσο θεωρώ ότι το δωρεάν θα βοηθήσει τους καταναλωτές και κυρίως τους καταναλωτές οι οποίοι ε, δεν έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ε, θεωρώ ότι το ADR είναι εξαιρετικά χρήσιμος μηχανισμός αλλά παράλληλα νομίζω ότι για την στήριξη αυτού του μηχανισμού πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και οι συλλογικές προσφυγές. Βλέπω την αγωνία του Προέδρου και βάζω μία τελεία εδώ, επιφυλάσσομαι για την ε, επόμενη έκθεση. Thank ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Ρούσο. δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ίσως μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια. και μετά και στον κύριο Άλεμπερτ τον, από την εταιρεία, αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Πρώτα, κυρία Ρούσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί πράγματι δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεβέλτ για την παρουσίαση της έκθεσης η οποία έκθεση βασίζεται ε, σε δουλειά που έχει γίνει ήδη για μας για την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ πέρυσι. Απλά εμβαθύνει, η παρουσίαση αυτή στην ανάλυση που σας ανέφερα. Ε, τώρα, όσον αφορά την ανάγκη να υπάρχει ένα νομικό εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προβάλλεται ε, και για εθνικές ε, διαδικασίες επίλυσης διαφορών και για διασυνοριακές. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην έκθεση του κυρίου, του κυρίου Ροσφό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ροσφό για τη δουλειά του. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή ε, ευθυγραμμίζεται με αυτά τα οποία προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε επιβεβαιώνω ότι ε, θα υποβάλουμε πρόταση οδηγίας για τα ADR. Θα σκεφτούμε και το όνομα, τον τίτλο. Ε, θα πρέπει ο τίτλος να είναι και νομικά βιώσιμος. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο, το, την ονομασία των συστημάτων, αλλά θα το δούμε. Στην πρόταση αυτή οδηγίας ε, ε, θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη. Συνεπώς, δεν θα θέσουμε στο περιθώριο αυτό που ήδη λειτουργεί στα κράτη-μέλη. Θέλουμε απλώς να καλύψουμε τα κενά. Δηλαδή ε, τα ADR να φτάσουν και στους τομείς και στις περιοχές στις οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμα. Και πάλι ε, βρισκόμαστε στην ίδια συχνότητα με τους ηγητές. Τώρα σε ό,τι αφορά την χάρτα ε, για τις αρχές των συστημάτων ADR ε, θα το σκεφτούμε ως συμπληρωματικό στοιχείο του νομοθετικού κειμένου κάτι δηλαδή που θα υπογραμμίζει τις αρχές των ADR που έτσι και αλλιώς θα συμπεριλάβουμε στο νομοθετικό μας κείμενο. Σε ό,τι αφορά τις ίδιες αυτές τις αρχές, συμφωνούμε με την απαρίθμηση που γίνεται στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά τον, χαρακ... τον δωρεάν χαρακτήρα για τους καταναλωτές, ε, ακούσαμε και τις παρατηρήσεις του κ. Μάγερ και της κ. Βάιλερ και της κ. Ράπτη Πιστεύουμε και εμείς ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την, ε, το δωρεάν χαρακτηρίο του καταναλωτέ, αλλά θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να δεχτούμε ο καταναλωτή να φέρει ένα τμήμα του κόστους, ενδεχομένως συμβολικό, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση, κατάχρηση του συστήματος. Σχετικά με το θέμα που υπογραμμίζει ο κ. Ροσφόρ σε ό,τι αφορά το είδος των, ε, ε, των ε, υποθέσεων θα πρέπει να και συμφωνούμε και εμεί ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στις C2B, δηλαδή ε, θέματα καταναλωτών, ε, καταναλωτών εναντίον επιχειρήσεων. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαμεθοριακές ε, διαφορέ, πράγματι θα μπορούσαμε να έχουμε μια, μια ιστοσελίδα χωρίς να δημιουργήσουμε μια καινούργια δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιπλέον των εθνικών δομών. Η ιδέα είναι να έχουμε μια online πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών που θα καλύπτει τις διαμεσοριακές ε, διαφορές και θα είναι μια πλατφόρμα ε, που θα διευκολύνει την διασύνδεση των ADR σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η πλατφόρμα θα βασιστεί ενδεχομένως σε εμπειρίες που έχουμε ήδη από το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή και θα αποτελέσει μια ενιαία θηρίδα για όλους τους καταναλωτές ε, ε, που θα παραπέμπει τον καταναλωτή στην αντίστοιχη αρμόδια, στο αντίστοιχο αρμόδιο εθνικό EDR. Επίσης, ε, η Κομισιόν έχει την πρόθεση να υιοθετήσει μια πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία μιας ε, πλατφόρμας online για την επίλυση διαφορών ε, παράλληλα με την πρόταση που θα υποβάλουμε για τα πρόταση οδηγίας που θα υποβάλουμε για τα ADR. Είναι πολύ σημαντική επίσης η ενημέρωση του κοινού, θα έχουμε, πρέπει να, έχουμε, να υποβάλουμε ε, προτάσεις και για το θέμα της ενημέρωσης του καταναλωτή. Έχουμε βάση δεδομένων στην Κομισιόν, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με αυτό. Η δική μας ε, βάση δεδομένων κάνει απλώς μια καταγραφή ε, ονομαστική καταγραφή των ε, ADR που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το σήμα ποιότητας, ε, είναι ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα το σκεφτούμε, θα το λάβουμε υπόψη. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, συλλογικές προσφυγές, λαμβάνω υπόψη τα σχόλια όλων των ομιλητών και την συζήτηση που θα λάβει η χώρα εν ώψη του επόμενου σημείου της ημερησίας διάταξης θα σας αναφέρω τα σχόλιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ε, διευκρινίσατε τα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Είναι σαφής η στρατηγική σημασία του όλου θέματος και θέλω να απογραμμίσω ότι εδώ πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που συμφώνησε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την επίλυση των διαφορών για τους καταναλωτές να είναι δικής μας αρμοδιότητας. Ε, και αυτό είναι σαφές όσον αφορά τη γνωμοδότηση που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο Κύριε Αλεβάρτε, ε, θέλετε να τοποθετηθείτε πολύ σύντομα σε συγκεκριμένα θέματα, γιατί ήθελα να δώσω μετά το λόγο στον κύριο Ροσφό. Ε, θα ήθελα πολύ σύντομα να σχολιάσω ε, κάποια θέματα που ετέθησαν και για τα οποία έχουμε στοιχεία. Το πρώτο ερώτημα που ετέθη είναι κατά πόσον υπάρχουν έρευνες για προγράμματα διαθέσεις διαφορών από πλευράς μεταξύ κράτους και επιχειρησεων b P2B. Ε, είναι λοιπόν θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων, όμως αφορά τους εμπειρογνώμονες και όχι τους ε, καταναλωτές. Και εάν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει signposting. Πράγματι, ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ε, χρειάζεται σε εθνικό επίπεδο. Το θέμα των αρμοδιοτήτων για την επίλυση διαφορών. Κοιτάξτε, όταν κάναμε έρευνες το 2009 ε, εκ μέρους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα του ε, διαμεσολαβητή του Ombudsman αυτό δεν τίθεται καν γιατί υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί ε, που μοιάζουν να λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν λοιπόν προδιαγραφές ε, στην σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι προδιαγραφέ αυτέ βέβαια δεν είναι πάρα πολύ πρακτικές, δεν εφαρμόζονται εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ αφηρημένες, ε, γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να έχουμε και πρακτικές ε, οδηγίες που βοηθούν στο πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά τα συστήματα. Πάντως το θέμα των αρμοδιοτήτων πράγματι αποσχολεί όλους και τις επιχειρήσεις. Κατόπιν, τέτοιο ένα θέμα που αφορά στο κόστος. Προφανώς Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το κόστος και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα τα συστήματα έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Ε, σημασία έχει τα συστήματα να είναι εφαρμόσιμα. Αυτά είχα κατ' ουσία να απαντήσω. Και κάτι άλλο, το τελευταίο γιατί λέτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ε, νομικό εργαλείο. Πρώτον, πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχουν ε, προβλήματα σημαντικά για του καταναλωτέ. Σαφώ ναι, αυτό το σύστημα είναι χρήσιμο τη ε, επίλυση διαφορών. Λέμε ναι, και το τρίτο ερώτημα είναι κατά πόσον το σύστημα αυτό, το εναλλακτικό, θα εξελιχθεί περαιτέρω έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτή να βρει ένα παρεμφερέ σύστημα και σε άλλο κράτο μέλο. Από την εμπειρία μα των τελευταίων δέκα ετών, μπορώ να σα πω ότι κάτι τέτοια, δηλαδή ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εφόσον υπάρχει και η απαραίτητη νομοθεσία. Ο κύριο Ροσφόρ. Για να καταλήξει. Ναι, πολύ σύντομα. Τρία σχόλια. Ευχαριστώ τους Κιώδης και τους συναδέλφους που έκαναν τόσο επικοδομητικά σχόλια. Θα τα λάβω υπόψη μου. Τα τρία σημεία είναι το κόστος, οδηγία ή χάρτα και οι συλλογικές οργανώσεις. Λοιπόν, για το κόστος καταρχήν, όπως είπε ο κύριος Φόξ, ο δωρεάν χαρακτήρας είναι μεν βασικός, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της εναλλακτική επίλυσης διαφορών είναι να μην πάει κανείς στο δικαστήριο. Όταν πηγαίνει κανείς στο δικαστήριο για παραπτώματα είναι δωρεάν η διαδικασία. Αν λοιπόν έχει κόστος η εναλλακτική διαδικασία, έστω και αν είναι μικρό, ενώ το δικαστήριο είναι δωρεάν, είναι αποτρεπτικό. Δεν πρέπει να καταλήξουμε λοιπόν μέσω του κόστους να ξαναοδηγήσουμε τον κόσμο στα δικαστήρια. Δεύτερον, χάρτα ή οδηγία. Νομίζω ότι χρειάζεται οδηγία. Ορισμένοι συμφωνούν, ορισμένοι διαφωνούν. Εντάξει. Αλλά δεν βλέπω είναι ποιο είναι το πρόβλημα με τη χάρτα. Χάρτα είναι μια λέξη που αρέσει στους διαμεσολαβητάς. Και δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι που επιβαρύνει περισσότερο τα πράγματα. Και τρίτο σχόλιο, η σχέση με τη συλλογική σύμβαση ή τη συλλογική συμφωνία. Πολύ συχνά είναι ατομικές διαφορές εκείνες που καταλήγουν σε εναλλακτική επίλυση. Οι ατομικές λοιπόν διαφορές δεν ε, συνδέονται με τις συλλογικέ συμφωνίες ή συμβάσεις. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν οι ΕΔ ως όπλο κατά των συλλογικών προσφυγών. Δεν είναι το ένα αντί του άλλου. Ούτε πρέπει να πούμε στους καταναλωτές και καταναλώτριες θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία για να αποφύγετε τη συλλογική προσφυγή. Θα υπάρχει η συλλογική προσφυγή ως τελευταία δυνατότητα άμα δεν λειτουργήσει η εναλλακτική. Αλλά να μην μπερδεύουμε την ατομική με τη συλλογική προσφυγή. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ περιεκτικά όλα αυτά με την παρουσίαση και μετά τη συζήτηση. Κύριε Ροσφόρ, στις 31 Αυγούστου θα εξετάσουμε την έκθεσή σας. Περνάμε τώρα, να σας πω όμως πρώτα κάτι. Καθυστερούμε. Ναι, να ευχαριστήσω και τους συντάκτες της παρουσίασης Civic Consulting. Σας ευχαριστώ όλους σας. Λοιπόν, έχουμε μόνο 20 λεπτά τώρα για την κυρία Ράπτη, αλλά και μετά τις διακοπές θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Έχω ήδη τον κύριο Ζουβά, Κρόιτσμαν, Φορκ, Κάμβα, Λίπη. Πρέπει λοιπόν μέχρι τις 12 να το λήξουμε αυτό. Έχουμε και την αξιολόγηση της Κομισιόν για τις συμβάσεις πίστοσης. Θα κάνουμε τις παρουσιάσεις και ίσως τα σχόλια αργότερα. Θα είμαι αυστηρότατος. Κυρία Ράπτη, όσο περισσότερο μιλήσατε τόσο λιγότερο θα ακούσετε τους σκιώδεις σας. Αργανώστε το μεταξύ σας. Εν τω μεταξύ σας δίνω το λόγο για να παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσή σας. Το πήρα το μήνυμα κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ταχύτατη. Ε, λέω λοιπόν πρώτον ότι συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο σημείο της ομιλίας του κυρίου Ροσφόρ και το προσυπογράφω. Δεύτερον, το ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα και οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ζημιές και να μην λαμβάνουν ε, αποζημιώσεις έτσι όπως θα έπρεπε ε, τρίτον, λέω ότι η Επιτροπή καλό θα είναι να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία. Τέταρτον, τονίζω, υπογραμμίζω, σημειώνω, με άλλα λόγια δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, στο ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατόν η έγκαιρη επίλυση διαφορών και η προσφυγή στα δικαστήρια να είναι η έσχατη λύση. Τέλος, υποστηρίζω και, και αυτό το επισημαίνω ότι το δικαστήριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την απόφαση για το αν είναι ή δεν είναι παραδεκτή η αξίωση η εκπροσώπηση και ο έλεγχος στον τρόπο ενημέρωσης των καταναλωτών. Βάζω μια τελεία εδώ, μη χαίρεστε κύριε Πρόεδρε, δεν τελείωσα ακόμα, και μεταφέρω δύο σημεία από την ακρόαση στην οποία ήμουν στην Επιτροπή, την κυρίως Επιτροπή για το θέμα του Collective Redress, των νομικών θεμάτων. Στο hearing έγινε ε, πάρα πολύ ε, καθαρό Πρώτον, ότι όλοι θέλουμε να είμαστε μακριά από το σύστημα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, υπάρχει μία πραγματικά ε, πλατιά οπτική από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και από την Κομισιόν. Η κυρία Ρέντινγκ δεν μας έδωσε ε, συγκεκριμένα την διάθεσή της, την πρόθεσή της και λέω τη δική της γιατί ξέρουμε ότι ενώ εμπλέκονται και ο κύριος Αλμούνια και ο κύριος Νταλή ε, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο με κάποιο τρόπο τον έχει η κυρία Ρέντινγκ. Μας παρουσίασε, είναι ανοιχτή στα πάντα και ε, κατέληξε στο ότι οπωσδήποτε ως το τέλος του χρόνου θα υπάρχει ανακοινοθέν ωστόσο κλείνοντας θεωρώ πραγματικά ότι θα βοηθήσει την κουβέντα μας και τον προβληματισμό μας το να σας διαβάσω την πρόταση με την οποία κατέληξε ο εκπρόσωπος του European Justice Forum ο οποίος λέει με δύο κουβέντες In conclusion, let us rather use a new European model of individual and collective redress based on ADR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 Thank Σας κατευχαριστούμε κυρία Ράπτη για αυτήν τη σαφέστατη παρουσίαση. τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ράπτη, αν είμαστε υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικής προσφυγής, αυτό το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές και καταναλώτριες αλλά και τις επιχειρήσεις. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία συλλογικής προσφυγής και σήμερα μπορούν να αποτελέσουν δουρίους ύπους για όλες τις καταχρήσεις που αναφέρατε. Επομένως, για να προστατεύσουμε και τις επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Επιτρέψτε μου τώρα να επανέλθω σε ορισμένα σημεία του κειμένου σας. Πρώτον για το εύρος, το πεδίο εφαρμογής. Βεβαίως θα βασιστούμε στον καταναλωτή και την καταναλώτρια, αλλά μια στιγμή μιλάτε για τον πολίτη. Μήπως αυτό είναι κάποια ασάφεια να λέμε από τη μία πολίτης και από την άλλη καταναλωτής. Τρεις φορές αναφέρεστε στις σχέσεις επιχείρησης και επαγγελματιών. Τι ακριβώς εννοείτε, συμπεριλαμβάνετε και τις επιχειρήσεις στο σχέδιό σας των συλλογικής προσφυγής. Έπειτα, για τη βασική συζήτηση μεταξύ opt-in και opt-out. Η έκθεσή σας νομίζω ότι δεν παίρνει θέση σαφώς, ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου και η ανάλυση του αμερικανικού παραδείγματος, αν δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιες καταχρήσεις, νομίζω δείχνει ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε κάποια προτίμηση υπέρ του opt-in. Τρίτον, η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι βέβαια βασικό πράγμα για να αποφευχθούν καταχρήσεις. Ιδιαίτερα η χρηματοδότηση από τρίτους που επιτρέπεται στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια πηγή καταχρήσεων γνωστή. Ορισμένοι ειδικεύονται στη διαχείριση συλλογικών προσφυγών για τρίτους και στην πραγματικότητα πρόκειται για κατάχρηση. Τέταρτον, δεν αναφέρεστε και θα ήθελα ίσως να υπάρχει αυτό στην αρχή να πληρώνει ο χαμένος. Έπειτα η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων καταναλωτών και καταναλωτριών. Μήπως θα έπρεπε να μιλήσουμε εδώ και για τη δυνατότητα να υπάρξουν κριτήρια αναγνώρισης της αντιπροσωπευτικότητας οργανώσεων των καταναλωτών και καταναλωτριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης στη συζήτηση διαμεσολάβηση και συλλογική προσφυγή ίσως δεν τονίζεται παρκώς τη δυνατότητα να ενισχυθεί η διαμεσολάβηση γιατί η συλλογική προσφυγή πρέπει να είναι η τελευταία φάση άμα αποτύχει η διαμεσολάβηση. Τέλος, σημειώνω με ενδιαφέρον ότι παραπέμπεται στις στα πρόστιμα που δεν πρέπει να γίνονται δεκτά πανευρωπαϊκά διότι είναι και αυτό πηγή κατάχρησης των συλλογικών προσφυγών, πρόστιμα ή αποζημιώσεις. Αυτά είχα να σας πω και εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθειά σας, τη συλλογική μάλιστα προσπάθειά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, συμφωνώ και παυξάνω με αυτά που είπε ο πρόλαλή σα. Ε, γι' αυτό δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε. Η συνάδελφος ε, η κυρία Ράπτη είπε ότι οι καταναλωτέ δεν παίρνουν αυτό που θα έπρεπε να λάβουν. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχει το δυνατότητα τη συλλογική αγωγή και υπάρχουν και διαφορετικέ νοοτροπίε. Α πούμε, όταν συζητήσαμε για την οδηγία περί των δικαιωμάτων των καταναλωτών, διαπιστώσαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να λύσουμε όλα τα προβλήματα, τη διαφορετικέ νοοτροπίε ε, με μία και μόνο οδηγία. Να σα πω, κυρία Ράπτη, τι ισχύει στη Γερμανία. Κοιτάξτε, στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη ε, προστασία απέναντι στου ε, πολίτε. Έχουμε 22.000 το 2009 υποθέσεις στα αστικά δικαστήρια για κάτω από 300 ευρώ. Και Έχουμε επίσης ε, και πολύ σημαντική καταφυγή σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ότι οι πολίτε ε, στη δική μου τη χώρα έχουν ε, τη δυνατότητα όποτε το επιθυμούν να καταφύγουν σε διαδικασίε διευθέτηση αφορών. και δεν χρειάζονται καν αυτό το σύστημα τη εναλλακτική διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν α προσέξουμε να μην ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρα και δεν νομίζω ότι αν καταθέσουμε τροπολογίες ε, θα λύσουμε το πρόβλημα. Εσείς στο τέλος ε, παραθέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σημείωσα fits with the national system είπατε, ταιριάζει με το εθνικό σύστημα. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ε, ε, τον συντονισμό σε υπερεθνικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν γίνεται γιατί υπάρχουν τελείως διαφορετικές δομές. Παραδείγματος χάρη κατά την ακρόαση ακούσαμε, οι Ιταλοί νομίζω μας είπανε ότι πριν καταφύγει κανείς στο δικαστήριο με συλλογική αγωγή όχι, ε, πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσει τη φιλική διευθέτηση. Αναγκαστικά να πάει εκεί για να μπορεί να καταθέσει αγωγή. δεν ξέρω αν θέλουμε αυτό να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Βάιλερ, κουνάτε το κεφάλι. Αλλά βλέπετε βλέπετε πόσο ε, διαφορετικέ ε, είναι οι νοοτροπίε. Οι Εγγλέζοι, παραδείγματο χάρη, που έχουν τη δυνατότητα συλλογική αγωγή, τώρα θέλουν να επαναχωρήσουν και να περάσουν στο δικό μα ε, το γερμανικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν α τα αφήσουμε τα πράγματα ω έχουν. Α προσπαθήσουμε απλά να δώσουμε περισσότερε δυνατότητε πολίτε διασυνοριακά. Αυτό είναι το θέμα, το διασυνοριακό. Όλα τα άλλα οι νοοτροπίε να παραμείνουν. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Και ο κύριος Φόξ νομίζω ότι έχει να ε, τοποθετηθεί επί του θέματος. Ευχαριστώ κυρία Ράπτη για τη δουλειά σας ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Εσείς γνωρίζετε και νομίζω και οι συνάδελφοι γνωρίζουν από την πρώτη μου παρέμβαση επί του θέματος ότι εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι λάθος. Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο που ακολουθήσαμε και με την οδηγία ε, δικαιωμάτων καταναλωτή. Θα σέρνεται υπόθεση για ολόκληρα χρόνια, δεν θα υπάρχει συμφωνία και γι' αυτό λοιπόν η δική μου η πρόταση είναι ας το ξεχάσουμε τώρα. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Θα χάσουμε χρόνο, θα χάσουμε κόπο και μετά από τρία-τέσσερα χρόνια θα καταλήξει μια ιονή, ένας ιονή που δεν θα αρέσει κανένα. Καλύτερα να ξεχάσουμε το θέμα και να τον καταλήψουμε τώρα. Επειδή όμω, κυρία Ράπτη και Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν θα εγκαταλείψετε την όλη υπόθεση τώρα, επιτρέψτε μου να σας δώσω μία συμβουλή. Δηλαδή, στη γνωμοδότησή σας, παράγραφοι 9, 10, 11, 12, ισχυρές, ε, ε, ισχυρά μέτρα κατά της κατάχρησης που μπορεί να προκύψει. Θέλω να πω ότι αν συστήσετε ένα σύστημα συλλογικής αγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς θα προσφέρετε κίνητρα να προκύψει ένα σύστημα όπου οργανώσεις, φορείς θα ενθαρρύνουν την αντιδικία, θα διεκδικούν υψηλές αποζημιώσεις και στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές ε, θα θελήσουν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και θα αρχίσουν να εγείρουν αξιώσεις με αποτέλεσμα να προκύψει γραφειοκρατία. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας προτείνω να περιορίσετε τη δουλειά σας σε αρχές που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κάποιες συγκεκριμένε διατάξεις για κατάθεση λογικής αγωγής. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να συνενέσει ο δικαστής. Αν λοιπόν εσείς θέλετε να περιορίσετε τη γνωμοδότηση σε κάτι τόσο απλό, να πείτε δηλαδή απλά ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει σύστημα συλλογικής αγωγής αλλά εναπόκειται στο κράτος μέλος να βρει την, ε, το σύστημα που του ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση του νομικού συστήματος που σχεί. Αν το κάνετε αυτό θα είναι χρήσιμο, αλλά οτιδήποτε άλλο αμφίσιμο θα οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα. Κυρία Βάιλερ και μετά η κυρία Ρουσό και η κυρία Ράπτη. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν είναι καινούρια. Γνωρίζουμε ότι ε, προβάλλονται συνεχώς ε, τα ίδια επιχειρήματα υπέρ και κατά. Νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει η στιγμή μετά από 7-8 χρόνια συζήτησης να καταλήξουμε σε αυτό το πολιτικό θέμα. Και τελειώνοντας θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, η ε, ο οικονομικός ε, πολιτισμός στην Ευρώπη πράγματι συγκλίνει. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Υιοθετούμε ορισμένα πράγματα από άλλες χώρες. Υιοθετήσαμε πολλά από τις σκανδιναβικές χώρες για την ισότητα, ε, για την καταπολέμηση διακριτικών μεταχειρήσεων. Αυτά δεν τα ήξερε η Ισπανία πριν το κάνει Υπάρχει λοιπόν μια σύγκληση. Και ένα πράγμα είναι σαφές. Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε τίποτα από την Αμερική. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό οπλοστάσιο, πολλά πολιτικά συστήματα δικά μας και δεν χρειάζεται να να τα υιοθετήσουμε από την Αμερική. Και τώρα, σε αυτό το θέμα, στη συλλογική αγωγή, επειδή ε, ενδιαφέρεστε για κάποιους ε, ειδικού λόγους, ε, λέτε ας υιοθετήσουμε το πρότυπο της Αμερικής. Η Αμερική δεν είναι το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε τα δικά μας. Right. Um, no other want to... Δεν θέλει κανένα άλλο μέλο το λόγο. Ο λόγο στον κύριο Ρουσό, στην κυρία Ρουσό και μετά στην κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ο Επίτροπο Ντάλι μίλησε για αυτό το θέμα στι 26 Μαου και η Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ στι 25 Μαου. Είπε, κυρία Ρέντινγκ, ότι η Κομισιόν εξετάζει αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα τη διαβούλευση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω θέση για τα ζητήματα τα οποία εθίγησαν. Η Κομισιόν, όπω επαναλήθηκε σήμερα το πρωί στην ακρόαση τη Επιτροπή Τζούρι, θα υποβάλει μια ανακοίνωση πριν το τέλο του χρόνου για να ε, προχωρήσουμε. Ευχαριστώ την κυρία Ράπτη για τις προσπάθειές της να μας υποδείξει ένα δρόμο. Σε ό,τι δεν αφορά τον κύριο Ζουβάν, θα ήθελα να πω ότι οτιδήποτε κάνουμε σε επίπεδο βασίζεται στην ανάγκη να αποφύγουμε σαφέστατα οποιασδήποτε καταχρήσεις και για αυτόν τον λόγο θα προβλέψουμε τις, ε, τα κατάλληλα, το κατάλληλο σύστημα προστασίας. Σε ό,τι αφορά τους κ. Φόξ και Κρόσμαν, όπως αναφέρθηκε και στην διαβούλευση, η, οτιδήποτε κάνει η Κομισιόν θα κάνει σεβαστά τα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Αυτή είναι και η λογική της διαβούλευσης ό,τι κάνουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σέβεται τα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Θα, ακολουθήσουμε πολύ, θα παρακολουθήσουμε πολύ κοντά τι εξελίξει και θα επανέλθουμε με ένα ανακοινωθέν πριν το τέλο του χρόνου. Πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί μετά την υιοθέτηση της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρουσό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ όλο το πρωί. Κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι να πρωτοπώ τώρα. Ε, έχω ένα ερώτημα. Εσείς όλοι εδώ είστε παλιοί. Εγώ είμαι καινούρια. Και αισθάνομαι και λέω μήπως είμαι η κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος με τους λύκους και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ε, σκέφτομαι λοιπόν και λέω Ξεκινάω από τον κύριο Φόξ. Ο κύριος Φόξ ήταν καθαρός, ξεκάθαρος από την αρχή. Από την πρώτη φορά που κάναμε αυτή τη συζήτηση είπε collective redress, thank you, δεν θα πάρω. Τελείως. Ο κύριος Ζουβέν μου είχε δημιουργήσει ελπίδες. Όπως επίσης και ο κύριος Κρόιτσμαν στη σημερινή παρουσίαση μου δείξαν ένα άλλο πρόσωπο. Και οφείλω να είμαι ξεκάθαρη. Έκανα μία γνωμοδότηση η οποία με, με βασάνισε πολύ. Γιατί κάποιος μου είπε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι δεν θα τα παρατήσετε εσείς και η Επιτροπή. Εγώ ως άνθρωπος γενικά δεν τα παρατάω. Και Ίσως είμαι και λίγο συγκρουσιακός τύπος. Έτσι λοιπόν για να βγάλω κύριε Ζουβέν αυτήν τη γνωμοδότηση, την ε, πολύ έτσι light, παιδεύτηκα πολύ και συγκρούστηκα και με αρχές δικές μου προσωπικές, αλλά και με τα πιστεύω τη σοσιαλιστική ομάδας, του σοσιαλιστικού κόμματος στο οποίο ανήκω, αλλά και με τα πιστεύω που επικρατούν στην Ελλάδα θα ήθελα αυτό κάπου όλο αυτό που σας είπα να το βάλετε στην άκρη του μυαλού σας. Κατέληξα λοιπόν στο, ε, σε αυτήν τη γνωμοδότηση θέλοντας να αφήσω ανοιχτά όλα τα περιθώρια για συζήτηση. Γιατί πιστεύω ότι όταν ένα θέμα συζητείται επιμακρών, όπως αυτό, κάποια στιγμή έρχεται η φάση της ορίμανσης Είμαι αισιόδοξη, είμαι ε, ονειροπόλα. Θεωρώ ότι ίσως τώρα να είναι η πρώτη φάση της ορίμανσης. Έτσι λοιπόν κύριε Ζουβέν, σκοπίμως δεν αναφέρθηκα στο opt-in ή opt-out. Γιατί αν ερχόμουν εδώ με μια γνωμοδότηση που θα έλεγα ξεκάθαρα, κοιτάξτε να δείτε κύριε και κυρίες, εγώ θέλω opt-out, τελεία και παύλα. Αυτό είναι. Τότε για ποιο λόγο να κάναμε συζήτηση. Εγώ είμαι ανοιχτή, θέλω να ακούσω τα πάντα. Ε, χρηματοδότηση. Βάζω μερικές ιδέες. Να, η αρχή να πληρώνει ο χαμένος. Και εδώ συζητώ. Και εδώ συζητώ. Ε, τώρα, καταναλωτής, consumer, citizen. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια. Κάθε πολίτης είναι και καταναλωτής. Και υπάρχουν τρία στοιχεία επειδή θέσατε και το θέμα των επιχειρήσεων. Το είπα και στην προηγούμενη παρουσίαση. Στην Ελλάδα ο κορμός της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα έχω κάθε λόγο να τη σκέφτομαι. Στην Ευρώπη ο κορμός είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παύλα, καταναλωτές. Υπάρχει ο μεμονωμένος καταναλωτής και υπάρχουν και οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Και εδώ σκέφτομαι δύο πράγματα. Όταν μιλάμε για, τον καταναλωτή είναι σαν, σαν να μην το αναγνωρίζουμε όταν αγοράζει ένα προϊόν το τεκμήριο της αθωότητας τον αντιμετωπίζουμε ότι θα αγοράσω ένα κινητό τηλέφωνο και πίσω από το πρόσωπο αυτού που αγοράζει ένα κινητό τηλέφωνο ίσως είναι κάποιος πονηρός καταναλωτής που μπορεί και μόνος του να το ρίξει κάτω, να κάνει ζημιά και να προσφύγει στην Νόκια και να την κρεμίσει την Νόκια. Για όνομα του Θεού. Λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Υπάρχουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν στον κόσμο δουλειά έχουν χιλιάδες εργαζόμενους. Άρα δεν είμαι τρελή να θέλω αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις να τις δω να ζημιώνονται, διότι αν πέσουν τα κέρδη τους, αν σταματήσει η δραστηριότητά τους, θα βρεθούν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Ε, χρησιμοποιώ ακραία παραδείγματα γιατί θέλω πραγματικά να σας πείσω κύριε πρόεδρε επιτρέψτε μου δώστε μου λιγάκι χρόνο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο θέλω να σας πείσω πραγματικά για την ειλικρινή μου διάθεση να βρούμε ένα αυτό που λέτε εσείς εδώ και όταν ήρθα ηχούσε περίεργα στα αυτιά μου να βρούμε ένα καλό συμβιβασμό. Αν είναι να μην κάνουμε τίποτα, τότε πραγματικά δεν βλέπω το λόγο να, να συνεχίζεται αυτή η κουβέντα. Ε, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε και δεν θεωρώ, για παράδειγμα, ότι είναι το κομβικό σημείο το opt-in ή το opt-out δεν θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο σε αυτή την γνωμοδότηση τελικά και όχι έκθεση έχει σημασία το να υπερασπιστεί ο καθένας τα στενά κομματικά του συμφέροντα. Και σας λέω πραγματικά ότι για μένα ήταν θετική έκπληξη το γεγονός ότι στη σημερινή ακρόαση στην κυρίως Επιτροπή, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, το κλίμα ήταν πραγματικά, το υπογραμμίζω, τελείως διαφορετικό από αυτό που άκουσα εδώ. Υπήρχε από όλες τις πλευρές, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μία διάθεση να συζητήσουμε κοιτώντας προς το κέντρο του κύκλου της Ευρώπης και όχι προς την περιφέρεια. Και αυτό για μένα είναι ελπιδοφόρο για τους καταναλωτές πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για την Ευρώπη και συνολικά για το πολιτικό σύστημα αυτής της Υπήρου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κόντρα Αμερική-Ευρώπη υπάρχει και πάντα καλά κρατεί. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει τα φόντα, έχει τους ανθρώπους, έχει τα μυαλά να πάει ένα βήμα μπροστά. Εδώ βάζω τελεία κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ παθιασμένη η απάντησή σας. Πολύ καλή. Θα συνεργαστείτε βέβαια με τους σκιοσηγητές. Είσαστε οι συγγήτρια όλης της Επιτροπής, οπότε ε, ελπίζω ότι ε, θα βρείτε μια συμφωνία εκεί, ένα κοινό παρανομαστή και τελικά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Οι σκιώδεις έχουν μέχρι τις 19 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα να υποβάλουν τροπολογίες για να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ξανά στις 19 Σεπτεμβρίου. Και ελπίζω όλο αυτό το χρονικό διάστημα να τα βρείτε με τους ε, εισηγητές, με τους κοιόδης εισηγητές, συγγνώμη. Ε, ελπίζω ότι το, και οι, θερινοί, οι θερινές διακοπές να μας βοηθήσουν. Θα τα πούμε μετά τις διακοπές ξανά για αυτό το ζήτημα. Ε, έχουμε άλλη μια πρόταση να συζητήσουμε μια έκθεση για το θέμα των πιστοτικών συμφωνιών σχετικών με ε, την αγορά κατοικίας. Ε, σε συνεργασία με την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η σχέση μας με αυτήν την Επιτροπή είναι λίγο δύσκολη γιατί εξαιτίας της οδηγίας ε, ε, πιστώσεων στους καταναλωτές. Ε, και της ε, συνεργασίας μας ε, στο παρελθόν ξανασυζητάμε το θέμα των όρων με, με, σύμφωνα με τους συνεργαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε την έκθεση αυτή και την μελέτη επιπτώσεων. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αφιερώσουμε σε αυτό το ζήτημα τα επόμενα 25 λεπτά. Η ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή θα γίνει αργότερα, αλλά πιστεύω ότι αυτή η παρουσίαση της μελέτης επιπτώσεων ε, θα μας βοηθήσει Ο κ. Φιλίπ Πελέ ε, είναι εδώ και θα μας την παρουσιάσει. Έχουμε τις διαφάνειές σας. Θα μπορούσατε ε, σε 10 λεπτά να έχετε ολοκληρώσει. Ε, έχουμε και τους συγητές. Ο Κρόιτσμαν είναι εδώ. Ο κ. Φόξ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την μελέτη επιπτώσεων. Έχουμε αντίγραφα των διαφανειών σας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το πιο γρήγορο. Είχα υπολογίσει 30 λεπτά, τέλος πάντων. Για κάθε νομοθετική πρόταση ε, που υποβάλλει η Κομισιόν, ε, δημοσιεύει και μία ε μια μελέτη πτώσεων. Και σε αυτή την περίπτωση το ίδιο γίνεται. Ε, για αυτή την ε, περίπτωση ε, είχαμε μια πράσινη βίβλο το 2005, άσπρη λευκή βίβλο 2007 που επίσης συνοδεύτηκαν από μελέτες επιπτώσεων, διαβούλευση το 2009, ακρόαση το ίδιο χρόνο ε, νομοδότηση της ΕΟΚΕ και εκτενή συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε κάνει μελέτες, οφέλους ε, κόστους, έχουμε εξετάσει παραδείγματα το παρελθόν, έχουμε έρθει σε επαφή με οργανώσεις των, των καταναλωτών και του, το, του κλάδου. Όλα αυτά τα, όλο αυτό το υλικό μπορείτε να το βρείτε στο, στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Uh, ε, Ευτυχώ η, ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με τα στεγαστικά δάνεια που αντιμετώπισε η αμερικανική αγορά. Παρ' όλα αυτά έχουμε υψηλό επίπεδο ε, δανείων το 2008 το 10% ε, των οικοκυριών έχουν τέτοιου είδους δάνεια. Έχουμε αύξηση του ε, ποσοστού ε, αδυναμίας πληρωμής και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πολλές κατασχέσεις. Έχουμε ξεκινήσει εργασία στην Κομισιόν για να αποφύγουμε τέτοιου είδους κατασχέσεις. Παρ' όλα αυτά ε, έχουμε ε, σε πολλές χώρες ε, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε το 90% για παράδειγμα των δανείων να εκδίδονται σε ευρώ σε χώρες οι οποίες δεν είναι στη ζώνη του ευρώ Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ισοτιμίας ε, και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν υπάρχει σύστημα επίλυσης διαφορών ε, καθώς επίσης έχουμε και αύξηση του, σχέση της σχέσης δάνειο προς αξία σε πολλές χώρες. Ε, ε, έχουμε σε ορισμένες χώρες προβλήματα σε αγορές. Ε, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ε, διαφορά στην ενημέρωση του καταναλωτή σε πολλές χώρες οι καταναλωτέ δεν είναι ενημερωμένοι όταν λαμβάνουν ένα δάνειο, Καθώ επίσης έχουμε και διαφορά στα κίντρα που δίδονται ε, μέσω χαμηλών ε, επιτοκίων κλπ. Επίσης έχουμε προβλήματα και στις ρυθμιστικές αρχές, το στη ρύθμιση. Ε, ε, δεν έχουν όλες οι χώρες ε, καταγραφή των διαμεσολαβητών και των πρακτόρων. Ακόμα και εκεί όμως που υπάρχει καταγραφή, δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Συνεπώς η κατάσταση έχει πολλές όψεις, κάτι που, που αυξάνει τις αυθαιρεσίες. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά την ρύθμιση του τρόπου ε, ε λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπάρχει ένας ε, εθελοντικός διοντολογικός κώδικας που εφαρμόζεται όμως με διαφορετικό τρόπο στα κρατημέλη και σε διαφορετικό βαθμό. Ε, έχουμε την οδηγία παραπλανητικής διαφήμιση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκεί δεν αναφέρεται τίποτα ειδικό για τα στεγαστικά δάνεια ή για τις διαφημίσεις σχετικές. Ε, η οδηγία πιστώσεων στους πιστωτικών, ε, καταναλωτικών, καταναλωτικών δανείων επεκτάθηκε και με αυτόν τον τρόπο ε, καλύπτεται, καλύπτεται η Ευρωπαϊκή Επικράτη με διαφορετικό τρόπο από κράτος σε κράτος. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα ε, δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τις πληροφορίες που του δινόντουσαν και να αξιολογήσει ε, τις υποχρεώσεις που έκπταναν από τα δάνεια που έχουν λάβει. Οπότε πρέπει να γίνει δουλειά εκεί και για την ενημέρωση του καταναλωτή. Οι ε, δομές χρηματοδότησης των δανείων ε, είναι πιο συχνές στις ΗΠΑ από τις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, αλλά και πάλι έχουν σημαντική επίπτωση και σε περιπτώσεις απώλεια ζωής και σε περιπτώσεις ε, ε, απολύσεων. Επιπλέον έχουμε εξετάσει έξι προβλήματα. Η διαφήμιση δεν είναι πάντοτε ε, ή συγκρίσιμη. Έχουμε δει ενδείξεις τέτοιων περιπτώσεων που επηρεάζουν πιο πολύ χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά. Στην Πολωνία είχαμε προσφορές αστικών δανείων με επιτόκιο 0%. Μη ρεαλιστικό αλλού ε, είχαμε διαφημίσεις για πολύ χαμηλούς, ε, χαμηλά επιτόκια που δεν ήταν όμως διαθέσιμα για το μέσο καταναλωτή κλπ. λοιπά. Ε, ε, πληροφόρηση επίσης ε, που δίδεται στους κανόνες δεν είναι επαρκής και καθαρή. υπάρχει οδηγία βέβαια, αλλά δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού και στον ίδιο βαθμό οι μεθοδολογίες για το ετήσιο ε, επιτόκιο ε, προβλέπονται επίσης από, κοινοτικό, από, τα την κοινωτική νομοθεσία αλλά ε, διαφέρει πάρα πολύ, διαφέρουν πάρα πολύ, διαφέρει πολύ ο τρόπος παρουσίασής τους και αυτό δημιουργεί προβλήματα στους καταναλωτές. συμβουλές δεν ήταν ε, επαρκείς πολλές φορές. Καθώς επίσης και βρήκαμε ότι σε κράτη με τα οποία έχουν κανόνες για την ε, συμβουλή, για την ε, χωρίς συμβουλών, ε, ε, οι καταναλωτές πιο εύκολα κατέφευγαν σε διαμεσολαβητή για να ζητήσουν αποζημίωση όταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ε, δεν είναι επαρκείς οι μελέτες ε, αξιολόγησης ε, της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. Οι περισσότεροι πιστωτές είναι, δρούν βέβαια νόμιμα, αλλά όχι όλοι. Δεν έχουν πολλές φορές επίσης αρκετές πληροφορίες για την διαμεσοριακή ε, δεν έχουν αρκετή πρόσβαση στις διασυνοριακή πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα. Επίσης δεν έχουμε επαρκή καταγραφή των διαμεσολευτών, των ενδιάμεσων της αλυσίδας ε, ε, χορήγησης δανείων Οπότε είναι πολύ δύσκολο κιόλα να, να επιβάλλουμε και ποινέ ή κυρώσει. Χρειάζεται επίση να καταγραφούν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα. Εκεί όπου υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, στο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε και την επαγγελματική κινητικότητα ε, των πρακτόρων μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επίσης δίνουν ε, στεγαστικά δάνεια χωρίς ε, άδεια σε έξι και αυτό αποτελεί ένα κενό του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες, έχουμε μακροοικονομικές συνέπειες ε, σε όλη την οικονομία γιατί ο δανεισμός γίνεται με τρόπο ανεύθυνο πολλές φορές ε, αυτό δημιουργεί οικονομική ασάφεια, ανασφάλεια και ε, μπορεί να οδηγήσει και σε σχέδια ε, προγράμματα σωτηρίας, διάσωσης όπως στην Ιρλανδία, στη Λετωνία κλπ. Επίσης υπάρχουν προβλήματα όταν τα αγαθά, τα κίνητα τα οποία πολλούνται δεν είναι κατάλληλα και ε, ε, καθώς επίσης και προβλήματα με, την, με υψηλούς δείκτες αδυναμίας πληρωμών. Κύριε Πελέ, θα πρέπει να σας ε, ζητήσω να βιαστείτε. Ε, είσαστε στο μέσο της έκθεσής σας και ακόμα και είμαστε στις 12 και 20. Από, ας περάσουμε στο, στην ε, διαφάνεια παριθμών 9. Ζητούμε, ε, ε, προτείνουμε μια, την υιοθέτηση μιας οδηγίας. Το καλύτερο θα ήταν να έχουμε ειδικές δικούς κανόνες για τις διαφημίσεις και το διαφημιστικό υλικό, την παρουσίασή του, ειδικού κανόνες για τις πληροφορίες που δίνουν τους την πρώτης υπογραφής, ε, ειδικούς κανόνες για τον υπολογισμό ε, της αιτήσιας ε, δόσης και του επιτοκίου, κανόνες για τις συμβουλές και τις εξηγήσει, για την πολιτική αμοιβή, τη δυνατότητα του δανειολήπτη να αρνηθεί συγγνώμη, του πιστωτή να αρνηθεί ε, το δάνειο αν η μελέτη ε, ε είναι αρνητική. Για τους ενδιάμεσους και τις, τα μη χρησιμοποιητικά ιδρύματα χρειαζόμαστε καταγραφή, αδειοδότηση ε, και επιτήρησή τους. Σε ό,τι αφορά το κόστος, τα κόστη ε, υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων κλπ. Ε, αλλά συνυπολογίζονται τα, οι δαπάνες μηχανογράφησης ε, και οι δαπάνες ε, που αφορούν τον ε, χρόνο που δίδεται, που αφιερώνεται σε συμβουλευτικέ υπηρεσίε. όλα αυτά τα μέτρα που προτείνουμε μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των ετοιμάτων δανείων. Αυτό όμως αφορά ε, τα μικρότερα εισοδήματα, αλλά δεν θα αποτελέσει κάτι τέτοιο πρόβλημα για όλη την κοινωνία. Γιατί θα με την ε, μείωση αυτή της προσφυγής σε δάνεια ε, ενδεχομένως θα μειωθούν και όλα τα προβλήματα στην οικονομία γιατί θα έχουμε λιγότερες περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής των δανείων. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ. Για τα ωφέλη να πω ότι ε, κάνουμε μια εκτίμηση, μια εκτίμηση μόνο. Ε, ε, αν, τα ωφέλη ανέρχονται από 1,2 σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. το κόστος για τον τομέα είναι από 383-622 εκατομμύρια για τα κράτη-μέλη και τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα, πιστεύουμε ότι ε, αναλύσαμε όλες τις αναλυτικές λύσεις και το καλύτερο είναι μια πρόταση οδηγίας και όχι αυτορύθμιση. Ω προ τα συμπεράσματα, όπω σα είπα, προτείνουμε την υιοθέτηση μια οδηγία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω, Πρόεδρε. Θέλετε να συνεχίσετε. Προτείνουμε λοιπόν μια οδηγία, αναφερόμαστε στο περιεχόμενό της. Η αξιολόγηση αντικτύπου ε, είναι 30 σελίδες και 300 σελίδες ε, ε, παραρτήματα θα τη βρείτε στο site μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά από τις συνεννοήσεις μας με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή κατάλαβα ότι το θέμα είναι ο διακανονισμός ή τη ευθέτηση της συμπεριφοράς της αγοράς αυτής, αλλά εσείς μιλήσατε μόνο για θέματα καταναλωτών και καταναλωτριών. Μας δώσατε χρήσιμες πληροφορίες και φαντάζομαι ότι, επιβεβαιώστε το μου, ότι την ίδια παρουσίαση θα είχατε κάνει και στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Τονίσατε δηλαδή το γενικό πλαίσιο. Αφού όμω ακόμη δεν συνεννοηθήκαμε με τη γραμματεία της Οικονομικής Ενωτική Επιτροπής, εντάξει, λοιπόν τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις, διότι δεν θέλω να εκμεταλλευτούμε πάλι τους ερμηνευτάς όπως εχθές. Έχω λοιπόν κάποιο χρόνο για σχόλια, σύντομα όμως. Μας δώσατε πολλές χρήσιμες πληροφορίες πάντως, θα τα ξαναδούμε ιδιαίτερα για την κοστολόγηση. Να ορίστε τι θα διαβάσετε στην παραλία συνάδελφοι. Ο κύριος Λέχνερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την ε, έκθεση. Θέλω μόνο να πω ότι το είπε και η Κομισιόν ε, στην αρχή ότι η κατάσταση στα κράτη-μέλη ποικίλει, διαφέρει πολύ όσον αφορά τα προβλήματα. Εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο να το λύσει κανείς με μια οριζόντια ρύθμιση, ούτε και νομοθετικά. Ε, δεν μπορεί κανείς διανόμου να επιβάλλει στο τέλος να αποπληρώνονται όλα τα δάνεια. Εγώ παρόλα αυτά ε, χαιρετίζω την προσέγγιση Κομισιόν ε, διότι ήταν αρκετά επιφυλακτική και διότι αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι αγορές αλλά οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολύ περιορισμένες. Θέλω να πω κάτι και για τους συναδέλφους που ενδεχομένως να μην το ξέρουν κύριε Πρόεδρε. Οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ήταν πάρα πολύ δύσκολες για να πω το λιγότερο. Όπως πολύ σωστά είπες η Επιτροπή αυτή έχει την άποψη ότι τα πάντα εμπλέκονται με τα χρηματοψηφιστικά και η μόνη αρμόδιοι είναι εκείνη αλλά εγώ θέλω να πω ότι τα πάντα δεν έχουν σχέση μόνο με τα οικονομικά αλλά και με τον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν με κνευρίζει πρέπει να πω το ότι ε, δεν ε, επιτύχαμε συμφωνία για το ότι για ορισμένα θέματα τουλάχιστον πρέπει να είμαστε αρμόδιοι και εμείς, να υπάρχει συναρμοδιότητα. Δεν θέλω να αναφερθώ με λεπτομέρειες αλλά θέλω να πω ότι ε, δεν θέλω να παραιτηθούμε από τις αρμόδιότητές μας. Ε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην είμαστε συναρμόδιοι και αυτό το θέμα να το υποβάλουμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί οι δύο εισηγητές ε, θα πρέπει να χάνουν δύο ώρες και αυτό δεν το λέω για λόγους ματαιοδοξίας. Δεν με ενδιαφέρει που είμαι εγώ εισηγητής, αλλά πρόκειται εδώ για την Επιτροπή και για τα δικαιώματα των συναδέλφων και πρόκειται και για το χρονοδιάγραμμα. Εγώ λοιπόν αμέσως μετά τις διακοπές ε, θα καταθέσω μια έκθεση, την έχω ήδη προετοιμάσει και είναι σχεδόν έτοιμη και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στην Επιτροπή οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν επ' αυτής, ε, γιατί υπάρχουν ε, δυσεπίλητα προβλήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και όσον αφορά τη διατύπωση και όσον αφορά το περιεχόμενο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε χρόνο. Ε, προς ενημέρωσή σας προβλέπετε στις 5 Οκτωβρίου να υποβληθεί σχέδιο έκθεσης που θα έχει μεταφραστεί εντωμεταξύ και τέλη Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε αν θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το Κοινοβούλιο να πρέπει μόνο του σε αυτήν την περίπτωση να θέσει όρια χρόνου και πίεση χρόνου. Αυτό αφορά τους ε, συναδέλφου ε, που ε, πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα. Αυτά ήθελα να πω σχετικά με την αρμοδιότητα επιτροπών. Και κάτι για τους αδέλφους που ενδεχομένω να μην το γνωρίζουν. Όπου υπάρχει συναρμοδιότητα με την ΕΚΟΝ, την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, ο κανονισμός προβλέπει έτσι και αλλιώ ότι η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή έχει την τελευταία λέξη. Αυτό απλά για να το ξέρουν μερικοί, για να γνωρίζουν ότι όπου είμαστε συναρμόδιοι και όπου επιθυμούμε τη συναρμοδιότητα γιατί προσκρούμε σε δυσκολίες. Παρακαλώ λοιπόν τη Γραμματεία σε αυτό το θέμα, ε, στην αρμοδιότητα να κάνει κάποιες έρευνες, να το κοιτάξει λίγο. Κατά τα άλλα, ε, την τελευταία φορά τοποθετήθηκα επί του θέματος και νομίζω ότι τώρα δεν έχει νόημα να ξαναμπούμε σε θέματα ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βανότ, έχετε κι εσείς να πείτε κάτι. πολύ σύντομα. Αναμένω την οδηγία για να σχολιάσω. Βέβαια όταν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μιλάει για ασυμμετρική πληροφόρηση προς ποια κατεύθυνση το εννοεί οι τράπεζες και τα πιστοτικά ιδρύματα δεν έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τους αιτητές δανείων ή οι καταναλωτές δεν έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται. Νομίζω και τα δύο. Καλό είναι να πληροφορήσουμε τους καταναλωτές, αλλά το βασικότερο όταν χορηγείται ένα δάνειο είναι για τα τραπεζικά ιδρύματα. Έχουμε διαφορετικά επίπεδα χρέωσης ανά χώρα. Στη Γαλλία η ιδιωτική χρέωση είναι ύψους του 60% ενώ στην Ισπανία 120% και η στρατηγική των τραπεζών παίζει και αυτή κάποιο ρόλο. Επομένως αυτή την οδηγία πρέπει να λέει κάτι για να πλαισιωθούν οι κίνδυνοι υπερβολικού δανεισμού. Την λεπτομερή αξιολόγηση θα τη δω στην παραλία όπως είπατε και εσείς πριν καταλήξω. Θα ήθελα όμως να δηλώσω προς την Κομισιόν ότι σημειώνω ότι το συνολικό κόστος που έχετε εδώ είναι 950 εκατομμύρια ευρώ ενώ κάτω κάτω στα έσοδα 1272 Επομένως είναι δαπανηρά αυτά τα μέτρα. Θα το ξαναδώ πιο προσεκτικά γιατί έχουμε δει πολλές φορές ευρωπαϊκή νομοθεσία να κοστίζει περισσότερο από ό,τι ωφελεί. Ευχαριστώ. Ωραία, έληξε ο χρόνος. Ευχαριστώ όλους όσους έμειναν μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φάση τώρα απλώς. Όσο για τις σχέσεις μας με την οίκον, θα συνεννοηθούμε και θα δούμε μετά τι έχουμε να πούμε. Πάντως σήμερα μας έδωσε πολύ περισσότερες πληροφορίες η Κομισιόν. Και νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο ότι μια από τι εναλλακτικέ λύσει που πρότεινε η Επιτροπή ήταν χρήσιμη για να δούμε ποια από τις επιτροπές είναι ακριβώς η αρμόδια. Πριν από 18 μήνες μας είχε πει προτείνει μια λύση την οποία δυστυχώς δεν δέχτηκε η Ένωση γιατί εγώ την έβρισκα πολύ οικονομική. Βλέποντας εδώ την πρόταση πρόκειται για σαφή εξέλιξη με βάση και αυτά που πάντοτε έλεγε η Επιτροπή μας. Βέβαια, οι σχέσεις μας με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή δεν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες μας. Και η κυρία Πόλτς και εγώ θα συμφωνούσαμε νομίζω από αυτό. Τις λεπτομέρειες συζητάμε τώρα, τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση και ευχαριστώ την Κομισιόν δεόντως και τον κύριο Πελέ για την προσέλευσή του. Δυστυχώς δεν είχαμε περισσότερο χρόνο να του δώσουμε, αλλά ήταν μια καλή αρχή. Τέλος. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι παραπάνω για τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες, προλαβαίνουμε ακόμη. Δεν νομίζω ότι στο Συμβούλιο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την οδηγία. Μερικές χώρες μέλη μάλιστα από ό,τι γνωρίζω δεν είναι και αθόλου ενθουσιασμένες. Είχατε πει κύριε Πελέ στην ανάλυση σας και στις διαφάνειές σας ότι άλλα ωφέλη όπως τα διαμεθοριακά τα έχετε σχεδόν πάλι στην άκρη. Αλλά το όλο θέμα των συζητήσεων μας με το Συμβούλιο ήταν ακριβώς εάν πρέπει να υπάρχει οδηγία που να μην λαμβάνει υπόψη της στα διαμεθοριακά. Αφού μας λέτε ότι το κύριο θέμα είναι η προστασία των καταναλωτριών και όχι τα διαμεθοριακά, αναρωτιέμαι, θα ξαναδώ τους αριθμούς σας για να δω μήπως η λύση που είχε προταθεί πριν 18 μήνες δεν είναι η πιο αποτελεσματική. Θα ξαναδούμε τους αριθμούς και μπορεί να χρειαστεί να σας ξανακαλέσουμε εδώ γιατί δεν προλάβαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και τους διερμηνευτές και διερμηνεύτρες που πάλι ξεπεράσαμε το χρόνο τους. Θα ξαναβρεθούμε στις 3 για να συζητήσουμε τα τυχηρά παιχνίδια. και παρακαλώ να είστε ακριβώς στις 4 και 20 εδώ γιατί θα έρθει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Πολωνίας. Καλή όρεξη λοιπόν.